Συνάδελφοι, παρακαλώ να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Καταρχάς, θα ήθελα να σας κάνω τις ανακοινώσεις μου σχετικά με τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. οι συντονιστές ε, συζήτησαν διάφορες ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λήφθησαν διάφορες αποφάσεις σχετικά με την ανακοίνωση της Κομισιόν για το πρόγραμμα Μάρκο Πόλο. Αποφάσισαν οι συντονιστές να προσκαλέσουν την Κομισιόν να παρουσιάσει την ανακοίνωσή της σε μελλοντική συνεδρίαση της Επιτροπής μας θεωρήθηκε ότι δεν χρειάζεται έκθεση αυτή τη στιγμή. Ωστόσο το πρόγραμμα Μάρκο Πόλο είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό αποφασίστηκε να έρθει εκπρόσωπος της Κομισιόν εδώ και να παρουσιάσει την ανακοίνωση. Για τα premium αποφασίστηκε ότι η Επιτροπή μας έχει συγκεκριμένη άποψη και θα πρέπει ο πρόεδρος της να διαβιβάσει επιστολή που θα αναφέρει τη γνώμη της Επιτροπής λόγω των χρονικών περιορισμών σχετικά με την έκθεση αυτή. Επομένως, ο πρόεδρος πρέπει να συντάξει επιστολή και άρα οι πράσινοι επανέρχονται στην κορυφή της λίστας για τις γνωμοδοτήσεις στο μέλλον. Γιατί πράσινη βίβλο για τις πολιτικές για το κλίμα και για την ενέργεια μέχρι το 2030, αλλά και για την έκθεση για την ηθαγένεια και για την έκθεση της ΕΟΚΕ και της Επιτροπής των Περιφερειών για το άρθρο 25 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η απόφαση των συντονιστών ήταν να μην ληφθεί η δράση. Επίσης, να μην ληφθεί η δράση και για άλλα έγγραφα συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για τον κανονισμό 33 του 2009. Η έκθεση για την πρόοδο των ανανεώσιμων και το έγγραφο εργασίας της Κομισιόν για το περιβάλλον των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο. Συγγνώμη γιατί έρχεται το τσάι και θέλω να βρω το φακελάκι που έχω και που προτιμώ. Συνεχίζω λέγοντας ότι επίσης δράση δεν θα αναλυφθεί ως προς το έγγραφο εργασίας που αναφέρεται στον οδηγό για την εφαρμογή ε, των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις, ούτε δράση θα αναλυφθεί για την κοινή έκθεση ως προς τη συμμόρφωση με τα κριτήρια ε, εισδοχής ε, όσον αφορά στη Σερβία. Η ειδική ομάδα για τον τουρισμό. Προβλέπουν οι συντονιστές έκθεση από τον κύριο Φιντάντσα και αποφασίστηκε να ξεκινήσει η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για το θέμα αυτό από το Σεπτέμβριο. Καλούνται όλα τα μέλη να υποβάλουν προτάσεις στους εμπειρογνώμονες μέσω της γραμματείας. Θα λάβετε λοιπόν ένα κάλεσμα από τη γραμματεία για να απαντήσετε και να συμβάλλετε στο θέμα αυτό. Τώρα, για το θέμα του καμποτάζ οι πράσινοι θέλησαν να τεθεί αυτό το θέμα και αποφασίσαμε, αποφάσισαν οι συντονιστές να καλέσουν τον Επίτροπο Σιμ για να το συζητήσουμε το θέμα αυτό μαζί του. Ως προς το 2014 τα project για τον προϋπολογισμό και τις προπαρασκευαστικές δράσεις αποφασίστηκε να εγκριθεί ο κατάλογος όλων αυτών των σχεδίων και να σταλεί στην Επιτροπή για συστάσεις πάντοτε περιλαμβάνοντας τα εφιστάμενα πιλωτικά προγράμματα. Αυτό ήταν η πρόταση της ηγήτριας κυρίας Ντυρά. Ως προς την επιτροπολογία, παρουσίαση δύο πράξεων κατά εξουσιοδότηση. Ο κύριος Ονίλ, διευθυντής της ε, ε, σχετικής γενικής διεύθυνσης, παρουσίασε δύο πράξεις κατά εξουσιοδότηση σε σχέση με το ITS μία για την οδική ασφάλεια, για την ε, καθολική πληροφόρηση, η άλλη για τα ε, ναρκωτικά και τα φάρμακα. Παρακαλώ ησυχία γιατί φαίνεται σαν να μπαίνετε σαν θεατές σε αγώνα ράγμπι, λέει ο πρόεδρος. Οι δύο νέες πράξεις εξουσιατότηση θα συμπεριληφθούν στην επιφυλίδα υπαριθμών 10. Υπό τα διάφορα οι σοσιαλιστές έθεσαν το θέμα της συγχώνευσης των αδειών οδήγηση και των διπλωμάτων οδήγηση και τη μεταρρύθμιση και τη οδηγία 126 του 2006, η συγκίτρια η κυρία Τικάου, η οποία θα υποβάλει τελικά έκθεση ζητώντας από την Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της γιατί ήδη περιλαμβάνονται αυτά στα του ταχογράφου. Αυτά λοιπόν για τη συνεδρίαση των συντονιστών. Έχετε απορίες, έχετε ερωτήσεις, σας ικανοποιούν οι πληροφορίες που σας έδωσα. Καλώς, τις δέχεστε. Χαίρομαι, περνούμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η ψηφοφορία. Έχετε όλοι τις κάρτες ψηφοφορίας σας. Okay, so just... Καλώς. Ε, να δώσω το λόγο στην κυρία Τικά. Δεχόμαστε λοιπόν ε, τα νεύματα. Να ε, κάνουμε μια δοκιμή παρακαλώ με τις κάρτες ψηφοφορίας. Ε, ξεκινάει η ψηφοφορία και έτσι έχω την ευκαιρία να πιω μια γουλιά τσάι όσο ψηφίζετε. Ψηφίσατε όλοι πόσα μέλη του ΕΛΚ, ίσως υπερβολικά πολλά αυτή τη φορά ή όχι κύριε Γραμματέα. Πέρα της ψηφοφορίας. Από ό,τι βλέπω όλοι συμμορφούνται με τους κανόνες προς στιγμή. Όλα κάποια πράγματα συμβαίνουν συνέχεια. Είναι γνωστά. Ξεκινούμε λοιπόν με την πρόταση για την Οδηγία Κοινοβουλίου και Συμβουλίου που τροποποιεί την Οδηγία 2009-16 για τον έλεγχο των κρατικών λιμένων. Εισηγητής ο υποφαινόμενος. 10 Απριλίου 2013. Να το κάνουμε δια της ηλεκτρονικής οδού. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Η κυρία Τικάου δίνει το σήμα. Ένας του ΕΛΚ παραπάνω. Γρήγορα, λίγο κράτησε το όνειρο. Ήταν πολύ καλό για να είναι αληθινό. Οι συντονιστές ίσως θα πρέπει να το εξετάσουν, ότι αν τρεις φορές γίνει αυτό, ε, την επόμενη συνεδρίαση να έχουν αποβληθεί για μία φορά. Πέρας της ψηφοφορίας. 37 υπέρ, ένας κατά, μη, καμία αποχή εγκρίνεται. Επόμενη ε, σχέδιο γνωμοδότησης. Συγγνώμη, έχετε δίκιο τηρετικά, 38. Ευχαριστούμε Σίλβια. Σχέδιο γνωμοδότησης για πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα φθοριούχα αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Με εισηγητή τον κύριο Παχνιό. Ξεκινάει η ψηφοφορία τροπολογία 40 υπέρ. Κατά αποχές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 Έστω. Νόμιζα ότι ήταν δικό μου το πρόβλημα. Ξεκινάει η ψηφοφορία για τη 46. Γι' αυτό πρέπει να το ελέγξω. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε την 47 δια της ηλεκτρονικής οδού. Ξεκινάει η ψηφοφορία, νομίζω ότι είναι η ίδια η πλειοψηφία, αλλά τέλος πάντων. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πάμε τώρα 50, 51 και 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 11, 8, 9 υπέρ. Κατά. Άποχες. Το επαληθεύουμε δια της ηλεκτρονικής οδού. Ξεκινάει ψηφοφορία ηλεκτρονική για 11, 8 και 9 μαζί.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 κατά αποχές να ελέγξουμε δια της ηλεκτρονικής οδού ξεκινάει η ψηφοφορία ηλεκτρονική για την 16. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. 17 υπέρ. 17 υπέρ λέει ο πρόεδρος. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 61 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται άρα η 18 καταπίπτει. Πάμε στην 70. Τεχνική σημείωση. Να τη διαβάσετε. Ποιος είναι υπέρ της 70. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται λόγω ισοπαλίας. 71 υπέρ. Κατά ε, αποχές. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Μήπως είναι το ίδιο. Ξεκινά η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. Άποχες. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά θα το ελέγξουμε. Ξεκινάει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά. Άποχες. Το επαληθεύουμε. Νομίζω ότι με την ίδια πλειοψηφία θα είναι το αποτέλεσμα. Όχι, όχι, εγκρίνεται, συγγνώμη, υπάρχει αλλαγή, εγκρίνεται η τροπολογία αυτή. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην 83. Υπέρ. Κατά. Αποχές θα το επαληθεύσουμε. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το επαληθεύσουμε. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την 83. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται πράγματι. 84 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 85. Καταπίπτει. Πάμε στην 86 υπέρ. Κατά. Αποχές να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Για την 86 ξεκινά ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 20 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21 του εισηγητή. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μπορώ και να το ελέγξω ηλεκτρονικά, αλλά και οι φιλελεύθεροι και οι σοσιαλιστές την υπερψήφισαν. Έστω, για την 21 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 87 υπέρ. κατά, αποχές, νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά θα το ελέγξουμε. Ξεκινάει η ψηφοφορία, ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας, απορρίπτεται. 88 υπέρ, κατά. Ξανά ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ για την 88. Κατά. Αποχές και θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικώς για άλλη μια φορά. Χαίρομαι που δεν προεδρεύω της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Το ελέγχουμε. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά εν πάση ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 89. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Ισοπαλία. Άρα απορρίπτεται. Ε, 90 τροπολογία μαζί με την τεχνική σημείωση. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές θα το ελέγξουμε δια της ηλεκτρονικής οδού. Ψηφίζουμε την 90. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμό 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 95. Του κυρίου Τέιλορ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές, θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία 97. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πέρα τη ψηφοφορία. Πράγματι εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά την 98. Νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά θα το εξακριβώσουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται πράγματι. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. τόσες πολλές τροπολογίες για μια γνωμοδότηση. Είναι γελίο, λέει ο πρόεδρος. Εκατό υπέρ κατά άποχες νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά ας το επαληθεύσουμε γιατί επέρχεται η κόποση της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι για την 100. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6. Καταπίπτει. Όχι, δεν καταπίπτει. Ζει και βασιλεύει. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 3. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 116 της κυρίας Wills με την τεχνική σημείωση. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, το ελέγχουμε ηλεκτρονικός. 117 ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίες Εγκρίνεται. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 115. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 128 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 122 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά να δούμε την τροπολογία 118. Ξεκινάει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. 119. Ξεκινά η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 45 είναι η επόμενη. Όχι, καταπίπτη. Ως γνωστόν. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές θα το επαληθεύσουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 27. Υποπτεύομαι ότι έχει απορριφθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Πράγματι απορρίφθηκε. 28 υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται με την ίδια πλειοψηφία. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 127 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 1 την προφορική για το εκτιμώντας 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ξανά, η τροπολογία 1 υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία υπαριθμών 1. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι είναι η ίδια πλειοψηφία, αλλά θα το επαληθεύσουμε. Συγγνώμη που ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τόσες πολλές φορές, για δύο-τρεις τροπολογίες είναι μόνο το θέμα. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται σαφέστατα. Η τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές και αυτό το επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά θέλω να είμαι σίγουρος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ξεκινά η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 29 υπέρ, 12 κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια κύριε Παχνιού. αλλαγή βάρδιας. Πάμε τώρα στην γαλάζια ανάπτυξη του κυρίου Δανέλη. it's a bit more shaded, is it? Mm. So compromise one. 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19 με προφορική τροπολογία. Υπάρχει ένσταση κατά της προφορικής τροπολογίας. Όχι, με την προφορική λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά αποχές επαλήθευση της 25 αρχίζει η ψηφοφορία ψηφίσατε τέλος εγκρίνεται λοιπόν 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται και αυτή. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 4 ως προσθήκη το πρώτο μέρος στην 35 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 38 προσθήκη στην 39. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε την 38. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές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 μόνο με τις λέξεις for example, for tax advantage, for ή e- Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 53 με την προφορική τροπολογία. Εκτός αν υπάρχουν ενστάσεις, όχι, ψηφοφορία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές παρακαλώ ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει νομίζω ότι εγκρίνεται ψηφίσατε όλες και όλοι τέλος α λάθος απορρίπτεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Από την αλία η 6 εκτός από τις λέξεις as well και τα λοιπά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές παρακαλώ ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει η ψηφοφορία ψηφίσατε τέλος και όντως εγκρίθηκε 67 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέτζι 11 εκτός από τα λόγια points out that κτλ. Τα βλέπετε στο έγγραφό σας. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 72 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 73 ως προσθήκη στην 72 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 9α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 75 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα, κατά τμήματα για την 76. Πρώτο τμήμα, <coughs> emphasize the need και τα λοιπά, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, advocates και επόμενα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και αυτό. Reggie 9, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 83 ως προσθήκη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση 84 αρχίζει η ψηφοφορία καλά τα πάμε αλλά νομίζω αρχίζει και σημειώνεται μια κόποση και δεν σηκώνουν όλοι καλά τα χέρια τέλος Απορρίφθηκε. Θέλατε επαλήθευση κύριε Γκρός για την 83 ε, έτσι δεν είναι. Μπορούμε να κάνουμε. Αν συμφωνείτε όλοι. Αρχίζει η ψηφοφορία λοιπόν. Επαλήθευση της 83. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται ας Κάνουμε την επαλήθευση. Αρχίζει. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 108 ε, υπέρ, κατά, αποχές. Επαλήθευση παρακαλώ, αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται. 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 113 με προφορική τροπολογία. Ενστάσεις, εάν όχι, με την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 113 εκπίπτει 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 115 είναι μόνο γλωσσικού χαρακτήρα αλία 1 μόνο το πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ψάρια 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά αποχές η ηλεκτρονική επαλήθευση, αν και νομίζω ότι απορρίπτεται, αρχίζει η ψήφος. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος και απορρίπτεται. Ρέτζι 7 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 118 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ, κατά, αποχές. Ας επαληθεύσουμε. 119 αρχίζει. Ψηφίσατε, τέλος. Απορρίπτεται. 120 υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. 121 είναι γλωσσικού μόνο χαρακτήρα. Φυσ 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται και αυτή. 124 είναι κατά τμήματα. Πρώτο χωρίς τις λέξεις του apply the precaution κτλ. Και το άλλο με. Ναι. Τώρα λοιπόν πρώτα χωρίς υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρα υποθέτω ότι το δεύτερο εκπίπτει, είναι. Α, πρέπει να το ψηφίσουμε λέτε. Καλά λοιπόν. <laughs> Ό,τι μου πείτε. Καλά, καλά. Υπέρ λοιπόν. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. <laughs> Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς ψηφίσαμε ψηφίσαμε να αφαιρέσουμε το precautionary principle και μετά ψηφίσαμε να το εντάξουμε πάλι. Ρέτζι 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 126. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 127. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 128 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα calls on the commission μέχρι microorganisms. Ζητεί από την Επιτροπή και άλλους μικροοργανισμούς, ας πούμε έτσι. Δεν, δεν είναι αυτός ο λόγος. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Ψέφι υπέρ των μικροοργανισμών. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο, and to employ the management, χωρίς τις τελείες βέβαια. Υπέρ, κατά, αποχές. Δεύτερο τμήμα λοιπόν, ξαναλέω, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 131 υπέρ, κατά, αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται ας κάνουμε την επαλήθευση ωστόσο ψηφίσατε τέλος εγκρίνεται τώρα αιτιολογικέ σκέψει τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχέ. εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές παρακαλώ επαλήθευση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 με ναι, ή χωρί μικροοργανισμού όπω θέλετε. Ψηφίσατε πέρας 38 υπέρ 5 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν και συγχαρητήρια στον κύριο Δανέλη. Κυρία Μάισνερ, μπορείτε να ψηφίσετε πρώτα την έκθεση της κυρία Σάβασα γιατί πρέπει να αποχωρήσει. Αν συμφωνείτε όλοι, ναι, προτιμάτε να <laughs> ψηφίσουμε την κυρία Σάβισαρ πρώτα. Δεν τους αρέσει γιατί είναι έτοιμα των φιλελεύθερων. Αλλά, μιας και είσαστε εσάς, δέχονται επειδή είστε εσείς. Να λοιπόν, πού είναι τώρα η έκθεση ή μάλλον η λίστα της κυρίας Έκθεση της κυρίας Σάβισαρ Πρόκειται για την τελευταία έκθεση. Την βρήκατε όλοι. Αρχίζουμε λοιπόν. Συμβιβαστική 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1. Υπέρ. Α, εκπίβει αυτή λέτε. Ποιος έφτιαξε αυτή τις αποχρώσεις του γκρι εδώ. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προχωρούμε στην 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές μάλλον όχι ακόμα επαλήθευση αρχίζει η ψηφοφορία ψηφίσατε όλες και όλοι πέρας απερευθεί 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 εκπίπτει 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση σημαντική 4 αρχίζει ψηφίσατε όλοι τέλος απερίφθη Εφτά τώρα, υπέρ. Υπέρ της 7, κατά. Αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση παρακαλώ της 9 αρχίζει ψηφίσατε τέλος εγκρίθηκε 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία αρχίζει η ηλεκτρονική δηλαδή ψηφίσατε πέρας 39 υπέρ 1 κατά και 0 αποχές συγχαρητήρια κυρία Σάβησαρα Ε, κάνουμε πάλι, πάλι εδώ την αλλαγή της βάρδιας στο προσωπικό έρχεται τώρα η ψηφοφορία κουν ούτε παραπάνω από 39 σελίδες δεν είναι παρά μια τεσσαράκοντα δηλαδή καλά λοιπόν Κύριε Κούν, όλοι έτοιμοι. Όλες και όλοι έτοιμοι να αρχίσουμε την ψηφοφορία της εκθέσεως Κούν. έκθεση του κυρίου Κούν για την καταλληλότητα των αυτοκινήτων, δηλαδή για την ε, καλή κατάσταση των αυτοκινήτων. Ε, καθόλου επίμαχο θέμα. Α, 20 σελίδες ψηφοφορίες. Είναι λίγο πολύ μαραθώνιος. Αρχίζουμε λοιπόν. Τροπολογίες 37 και 38 που ζητούν απόρριψη της πρώτης κομισιόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται.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 Κατά. Αποχές. Επαλήθευση παρακαλώ. 3α. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Μία παραπάνω ψήφο σημειώνεται εδώ του Λαϊκού Κόμματος. Τώρα εντάξει, τώρα έχει καλός, τώρα έχει καλός. Ωραία. Τέλος. Εγκρίνεται. Πού πάμε τώρα. 3β εκπίπτει, άρα συμβαστική 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 121 κοχ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 122 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ομοίως. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση λέει ο πρόεδρος 159. Α, όχι, λάθος. Συμβαστική 7. Συμβαστική 7. Επαλήθευση λοιπόν. Ψηφοφορία αρχίζει. Ψηφίσατε. Τέλος. Και εγκρίνεται. Η 174 εκπίπτει. Υπέρ. Μας μπέρδεψε ο πρόεδρος. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 31. Αυτή εκπίπτει ή καταπίπτει. Έτσι νομίζω ναι. «175 μπένιον» με τα λόγια «including examining the feasibility» κτλ. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 178 υπέρ, κατά αποχές επαλήθευση αρχίζει η ψηφοφορία ψηφίσατε πέρας εγκρίνεται 21 και 197 είναι ταυτόσιμες αυτές υπέρ, κατά, αποχές. Καλά, επαλήθευση λοιπόν. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. 207 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήμκο 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Τέλος. Και απερίφθη. 209. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 22. Α, μια στιγμή. Τότε που πήγαινε. Α, 179. 179. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελάτε ξανά μια φορά. Ξέρω ότι είναι κουραστική η ψηφοφορία. Σηκώστε καλά τα χέρια. 179. Υπέρ κατά αποχές έγκρινεται. Τώρα 23. 212-213, όλες μαζί αυτές, υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση, καλώς. Αρχίζει. Ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνονται. Καλά, τότε προχωρούμε στην 223. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Α, έχει αποσυρθεί. Τότε γιατί λοιπόν πιο βορέ κατά τμήματα αφού έχει αποσυρθεί το δεύτερο τμήμα. Καλά λοιπόν. 181. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. 181. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται. 224 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να δεν μπορούσε να σταθεί αυτό Δια... Α, συγγνώμη άρθρο 5 όλα είναι το ίδιο εκεί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνονται μάλλον οι 2.31 Εκπίπτει 2.32, 33, 37 και 22. Α, 2,32 και 2,33 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση, γιατί εγώ νομίζω ότι εγκρίνονται. Επαλήθευση λοιπόν αρχίζει. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνονται 37 και 22 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 238 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 239 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται ομοίως. Ήμκο 38 υπέρ. Κατά αποχές. Αποχές, 2.41 προφορική του κυρίου Φέρμπερ. Υπάρχουν ενστάσει, όχι, τότε λοιπόν τίθεται η ψηφοφορία με την προφορική. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 243 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ήμκο 41 υπέρ κατά επαλήθευση ύμκο 41 αρχίζει η ψηφοφορία ψηφίσατε τέλος απερίφθη Ήτρε 24 υπέρ κατά Επαλήθευση αρχίζει. Ψηφίσατε. Τέλος. Απερίφθη. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 45. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ας επαληθεύσουμε. 246 αρχίζει. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται λοιπόν. Ήμκο 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Η 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 Ακολουθεί λοιπόν η 2.49. Υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 250 υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 2.55 υπέρ. Α, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 2.56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ήτρε 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 268 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 269 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 278 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2,77 εκπίπτει. 2,80 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 281 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2,82 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έχουμε τώρα μια σειρά ταυτόσιμες τροπολογίες 35 μέχρι 308 υπέρ και 33 κατά αποχές εγκρίνονται. 306 εκπίπτει, 309 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 310 γλωσσική και η επόμενη. 316 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 314 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ...315 υπέρ... ...κατά... ...αποχές... ...εγκρίνεται... ...ΕΜΚΟ 59 υπέρ... ...κατά... ...αποχές... ...απορρίπτεται αυτή... 3, 18 και 19 είναι ταυτόσιμες, άρα ψηφίζονται μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 3, 20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3, 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρα εκπίπτει η 61. 3,25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3.27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.29 και 62 είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 3.30 και 63 το ίδιο υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 3.31 και 64 το ίδιο υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται και αυτές. 65 ΙΜΚΟ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκπίπτει 332. 3 33 και 66 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 3, 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αλληλούια, οι ρόδες μου δεν είναι αυτές. 3.35 Σερακιάνη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ήμουκο 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.37 του κ. Φέρβερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας κάνουμε παλήθευση. Συμβαστική 11 αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Συμβαστική 11 λοιπόν. Είστε όλοι ικανοποιημένοι και όλες. Ψηφίσατε πέρασε. Εγκρίνεται. Τρία σαράντα Ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές. Ναι, ας, ας κάνουμε καλύτερη επαλήθευση. Δεν είναι και τόσο σαφές το αποτέλεσμα. Ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν. Της κυρίας Ντυρόν ως προσθήκη η 345 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται με την ίδια ε, πλειοψηφία. Της ΙΜΚΟ εκπίπτει. 348 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 349 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.22 υπέρ κατά αποχές ας επαληθεύσουμε την 3.22 αρχίζει η ψηφοφορία Ψηφίσατε όλες και όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. Ακολουθεί ΙΜΚΟ 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3.23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3.53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3.24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ερχόμαστε στις αιτιολογικές σκέψεις, στα recital. Στο 3 έχουμε την τροπολογία 43 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 45 υπέρ, <clears throat> κατά, αποχές, εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΙΜΚΟ 2 εκπίπτει άρα 48 Φώστερ υπέρ κατά αποχές ας επαληθεύσουμε που νομίζω ότι εγκρίνεται 48 της κυρίας Φώστερ λοιπόν ψηφίσατε πέρας Α, ισοψηφία λοιπόν. Απορρίπτεται λόγω ισοψηφία. 44. Μπένιον υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 49. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, Απορρίπτεται. Ήμκο 3. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 50. Υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το ίδιο και 52. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 68. Αν με παρακολουθείτε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 ΙΜΚΟ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 και 75 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίζεται. Τέλος. Εγκρίνεται. 77 έτσι είναι. Ωραία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήμκο 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 89. Λάιχτφριντ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήμκο 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται και αυτή. Τελική ψηφοφορία. Αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. 33 ψήφοι υπέρ, 7 κατά και καμία αποχή. Τώρα, ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου. Αρχίζει. Ψηφίσατε. Τέλος. 32 υπέρ, 6 κατά και καμιά αποχή. Συγχαρητήρια για την έγκριση κύριε Κούν. Περνάμε τώρα στην κυρία Σενάλοβα. Ας προχωρήσουμε παρακαλώ με την έκθεση της κυρίας Συνάλοβα. Κύριε Πρόεδρε, πριν από το ξεκίνημα της ψηφοφορίας, ε, η 105 τροπολογία η δικιά μου θα ήθελα σας παρακαλώ να αποσυρθεί. Okay, thank you, Mr. Griesbeck. We will do that. Ευχαριστούμε. Θα το κάνουμε. Τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Να χρησιμοποιήσω το δικό σου έντυπο γιατί στο δικό μου δεν είναι καθόλου καλά σκιασμένες οι περιοχές, λέει ο πρόεδρος. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4 και 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβεβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προχωρούμε τώρα στο 2 υπέρ, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, αλλά θα το ελέγξουμε, ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος, εγκρίνεται. 59, 60, 61, 62 και 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. 53, 58, 64 μαζί. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 ψηφοφορία κατά τμήματα πρώτο τμήμα τεχνικές επιθεωρήσεις στην άκρη του δρόμου το δεύτερο αποσύρεται το πρώτο τμήμα ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική υπαριθμών 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά αποχές να το ελέγξουμε. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την 75. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στο τέταρτο μπλοκ τροπολογιών. 77, 78, 79 και 16. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 99 Γλωσσική. Πάμε στην 100. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 101. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 102. Υπέρ κατά. Αποχές. Να το επαληθεύσουμε γιατί δεν ψήφισε κανείς. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά τέλος πάντων. Ξεκινάει η ψηφοφορία ηλεκτρονική για την 102. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται πράγματι. Επέρχεται η κόποση της ψήφισης. 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 104 υπέρ κατά αποχές. Να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ξεκινάμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται. 107 υπέρ. Κατά αποχές να το ελέγξουμε. Νομίζω ότι εγκρίνεται, ξεκινούμε, εγκρίνεται, αλλά τέλος πάντων. Ξεκινούμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 107. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Πράγματι. Συμβιβαστική 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11 της Ήτρε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 117 ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές θα το ελέγξουμε. Θα το επαληθεύσουμε. Ξεκινά η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 119. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το επαληθεύσουμε. Ξεκινάει για την 122 η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται. Πάμε στην 121 της κυρίας Γκρίσμπεκ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 125. Διαγραφή. Ποιος είναι υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται, 126 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. 135. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 123 το πρώτο τμήμα γιατί το δεύτερο καταπίπτει πρώτο τμήμα του 123 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά ξεκινά η ηλεκτρονική ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρασε Απορρίπτεται. Πάμε στην επόμενη σελίδα. 141 είναι η επόμενη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 12. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη 13 της Ήτρε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 144 αποσύρθηκε. Όχι. Όχι. Ζει και βασιλεύει. 144. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Το επαληθεύουμε. Ξεκινάει για την 144 η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Μετά έχουμε αυτή που αποσύρεται. Πάμε στην 145. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 της Ήτρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 και 151 μαζί. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 152 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 153 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Στα παραρτήματα τώρα. 155 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 160 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 161 με την προφορική τροπολογία. Έχει κάποιος αντίρρηση στην προφορική τροπολογία. Όχι, τις ψηφίζουμε μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται μαζί με την προφορική τροπολογία. 1. Τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την 4. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρα η 50 καταπίπτει. Πάμε στη 47 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τελική ψηφοφορία. Ξεκινάει η ηλεκτρονική ψηφοφορία της νομοθετικής πρότασης. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 34 ψήφοι υπέρ. 5 κατά. Εγκρίνεται. Και για το νομοθετικό ψήφισμα ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. 32 υπέρ, 5 κατά. Καμία αποχή. Εγκρίνεται επίσης. Συγχαρητήρια στην κυρία Σενάλοβα και συγχαρητήρια στα μέλη που ήταν εδώ σήμερα και ψήφισαν. Επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, παρακαλώ. Έχουμε καθυστερήσει κατά 30 λεπτά. Θα το εκτιμούσε ιδιαίτερος να ε, δουλέψουμε λίγο πιο γρήγορα. Είναι εδώ ο κύριος Νταντά. Είναι ο συντάκτης της γνωμοδότησης. Όσοι είναι να φύγετε, φύγετε. Όσοι θα παραμείνετε στην αίθουσα, καθίστε για να προχωρήσουμε γρήγορα και να συζητήσουμε το θέμα που μας απασχολεί. Μία ολοκληρωμένη αγορά παράδοσης δεμάτων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Νταντά, Μπορείτε να ξεκινήσετε ήδη την παρέμβασή σας. Ας ελπίσουμε ότι θα σας ακούνε όλοι. Δεν μπορώ να περιμένω μέχρι να βγουν όλοι από την αίθουσα. Παρακαλώ μην μιλάτε στους διαδρόμους. Αποχωρήστε παρακαλώ. Πριν από 10 χρόνια αυτό το πράγμα η αγορά στο ίντερνετ ήταν μια εξαίρεση. Τώρα έχουμε 25% ε, θέσεις ε, αυτά τα τελευταία χρόνια. Αλλά αυτό εξαπλώνεται σε εθνικό επίπεδο. Τι βλέπουμε όμως ότι όταν περνάμε τα σύνορα τιμώ 9% των καταναλωτών, 18% των εμπόρων ακριβώς ε, είναι στο διαμεθοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Δεν είναι ότι ενοχλεί μόνο στις μεγάλες χώρες τους καταναλωτέ, αλλά και για τις ε, μικρότερες χώρες. Ε, και ε, αντί να αγοράζει εκεί, αγοράζει ένα προϊόν που έρχεται από την άλλη μεριά του κόσμου πολλές φορές ε, και εδώ κάθε επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου σε μια τοπική αγορά προσπαθεί στη συνέχεια να το κάνει και σε διεθνές επίπεδο. Αλλά υπάρχουν τις λειτουργίες διαθωτικές της αγοράς, το εμποδίζουν αυτό για την παράδοση αυτών των δεμάτων που είναι ιδιαίτερα περιπλοκή και η ποιότητα αυτής της υπηρεσίας είναι από τους κύριους παράγοντες για να πετύχει. Γιατί εάν δεν παραδοθεί όπως πρέπει ή είναι αλλοιωμένο τότε αποθαρρύνει τους αγοραστές και βέβαια υπάρχουν πολλά κενά, όπως σε διαμεθοριακό κυρίως επίπεδο η ευρωπαϊκή αγορά δεν είναι αγορά αυτή καθ' αυτή, είναι ε, σε διάφορα κομμάτια και διάφοροι ε, προσπαθούν να συνεργαστούν, ανταγωνίζονται όμως και έχουν θηγατρικές οι οποίες ε, επιδεινώνουν την κατάσταση και όχι μόνο αυτό που περιμένουμε μια κατάλληλη λειτουργία, η ποιότητα επηρεάζεται και πολλές φορές και η τιμή για την παράδοση είναι θόλη, δεν ξέρουμε ακριβώς. Ε, οι πρώτοι που υποφέρουν από αυτό είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν και τους περισσότερους που το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρώπη και δεν έχουν τα μέσα για να παρακάμψουν το πρόβλημα πέρα από αυτούς τους λίγους ε, ε, που είναι στην πρωτοπορία αυτού του ηλεκτρονικού εμπορίου που προσαρμόζονται γιατί είναι επιτόπου εκεί σε αυτή την αγορά για την παράδοση και προχωρούν ακόμα περισσότερο, πολύ περισσότερο γιατί οι ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις γίνονται και εξαρτώμενες από αυτούς. Λόγω της λειτουργίας και του ε, μικρού χαμηλού ανταγωνισμού, οι περισσότεροι από αυτούς που ασχολούνται με ηλεκτρονικό εμπορίο, οπωσδήποτε θα πρέπει να περάσουν από τους παραδοσιακούς που ασχολούνται με αυτό και πολλές φορές ε, δεν είναι γνωστή καθόλου ότι παρεμβαίνουν στην όλη διαδικασία και για την ανεχασιμότητα, για τις ετικέτες στην Ευρώπη. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι και να είναι ακριβώς η προσφορά της υπηρεσίας περισσότερο ατή και σε όλες τις περιπτώσεις ε, που θα πρέπει να έχουν τη μέση εθνικές αρχές να κάνουν να ασκούν ένα έλεγχο και να μπορούν να συνεργάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό ακριβώ χαίρομαι για την εργασία αυτών των ρυθμιστών των Ευρωπαίων για τις σταθεμικές υπηρεσίες που θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος τους. Και διαπιστώνουμε ότι ο καταναλωτής δεν είναι απόλυτα ελεύθερος για την επιλογή του, γιατί ο τρόπος επιλογής ε, προεπιλέγεται από αυτούς που ασχολούνται με το εμπόριο αυτό. Γι' αυτό ακριβώς ε, η ευθύνη να απέναντι στον καταναλωτή και για την όλη διαδικασία παράδοση θα πρέπει να τεθεί σαν θέμα και ακριβώς εκείνος είναι που θα ενημερώσει για αυτές οι υπηρεσίες που προσφέρονται για την όλη διαδικασία, την παράδοση όταν γίνεται η παραγγελία. Και πολλές φορές όμως αυτά τα πράγματα δεν είναι όπως πρέπει κατά τη διάρκεια τη παραγγελίας. Ε, Εκείνο θα πρέπει να παίξει επίσης το ρόλο των κατά κατάλληλο για ενημέρωση του για την εργασιμότητα κατά τη διάρκεια της πορείας ε, και να είναι ικανοποιητική για τον πελάτη που θέλει να ξέρει σε ποιο σημείο βρίσκεται το θέμα της παράδοσης. Ε, και ακριβώς θα πρέπει να υπάρξει ένας ένας χαρακτήρας αυτής της προφορίας ε, στις ιστοσελίδε για την αγορά. Εκείνα ακριβώ ακριβώς θα πρέπει να φέρουν σε πέρα στην καλή παράδοση η υπηρεσία, η αρμόδια για την επιστοποίηση κλπ. Και όλα αυτά θα πρέπει να αναγνωριστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο με διπλό θετικό για να βελτιώσουν εταιρείε αυτέ τι αποδόσει του για την παράδοση και ταυτόχρονα ο καταναλωτή να μπορεί να είναι σίγουρο για την αξιοπιστία αυτή τη υπηρεσία. Αυτά ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, αυτά τα κύρια που θα έπρεπε να έχουμε κατά νου. Ε, χρειαζόμαστε ένα καλύτερο ανταγωνισμό, καλύτερη ανεχνευσιμότητα και επίση να ξέρουμε ακριβώ ποιο είναι και πού υπεύθυνο. Ε, και τα χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε όλου να συνεργαστούν και η σχετική εμπορή και για τη σχετική διαδικασία παράδοσης ώστε η ευρωπαϊκή αγορά είναι περισσότερο αποτελεσματική και φθηνότερη και να επωφεληθούμε όπως πρέπει από το ηλεκτρονικό εμπόριο σε όλη την Ευρώπη. Δεν έχει οριμάσει ακόμα αυτή η αγορά και είναι πρόωρο να ε, νομοθετήσουμε σε αυτή τη φάση γιατί θα πρέπει ορισμένε απαντήσεις να δούμε πώς θα ε, έχουν χώρο σε μέσο πρόθεσμα στην αναθεώρηση της ταχυδρομικής οδηγίας. Θα σας δώσω αυτά σε λίγες ώρες και 5 ε, Σεπτεμβρίου θα το συζητήσουμε. Συνεργάστηκα πολύ καλά με τον εισηγητή της ΣΥΜΚΟ και συμμεριζόμαστε τις ίδιες απόψεις σχετικά με το θέμα. Thank you very much, Mr. I've got... Ευχαριστούμε πολύ κύριε Νταντέ, η κυρία Μάισνερ, Ζήλερ, Βίλς. Δεν έχει έρθει βέβαια ακόμα η κυρία Βίλς. Παρακαλώ να είστε όλοι ε, σύντομοι. Πρώτα η κυρία Βεθνιό, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μετά από τα συμπεράσματα του τον του συναδέλφου μου, η έποψή μου είναι ότι προδιαγράφεται μια θετική, πολύ καλή συζήτηση και πολύ καλή ε, συνεργασία για όφελος όλων. Και εγώ, σαν σκιοδησηγήτρια, ε, θα ήθελα να σας πω ορισμένα πράγματα που μας καθοδηγήσουν στη σκέψη μας. Αυτή η πράσινη βίβλος που παρουσιάστηκε στο τέλος πέρυσι από την Επιτροπή εγγράφεται στα πλαίσια της διάθεσης και την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη και μέρος της ε, πραξής ε, από τον Επίτροπο Μπαρνιέ το 2011 για το εμπόριο αυτό. Και αυτά τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει πολύ το εμπόριο, αλλά έχει ακόμα πολλές δυνατότητες ανάπτυξης, ε, κυρίως για τη δημιουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τύπη. Και επίσης αντιμετωπίζει όμως και προβλήματα, εμπόδια σχετικά με το διαμεθοριακό εμπόριο και είναι η γλωσσικά, τα γλωσσική φραγμή, η οργάνωση όσον, όσον αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών, τα διαφορετικά συστήματα πληρωμής και βέβαια το θέμα της παράδοσης. Η πράσινη αυτή βιβλίος προσφέρει λύσεις σε αυτό το τελευταίο σημείο που έχει διάφορες διαστάσεις. Ε, ακριβώς είναι μεταξύ και της ανάπτυξης ε, του εμπορίου και την ε, ενιαία διαδικασία, την ταχυδρομική και την όλη οργάνωση και καταλαβαίνουμε και γύρω-γύρω πώς επηρεάζονται τα πράγματα. Για αυτήν την πρώτη ανταλλαγή απόψεων να σας πω πώς ε, αναπτύσσονται ορισμένε σκέψεις απέναντι στον καταναλωτή πρώτα απ' όλα. Θεωρώ ότι είναι κάτι το πολύ σημαντικό να είμαστε βέβαιοι ότι κάθε βελτίωση της υπηρεσίας πάνω απ' όλα για την ταχύτητα αυτής της διαδικασίας ε, και της παράδοσης, πώς συλλέγονται τα πράγματα στα καταστήματα και αυτό το σύστημα να μην είναι μόνο να μην αφορούν μόνο μερικού. Θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουν να έχουν μια παρόμοια προσέγγιση όπως τη ταχυδρομική οδηγία, ε, ώστε να μην αγνοηθούν και οι αγροτικές ε, περιοχές ή ε, υπερπεριφερειακέ, οι μακρινέ. Και σχετικά με τον πρώτο λόγο που προκαλεί δυσπιστία για αυτή την, το είδο πώληση, δηλαδή κλοπή, καταστροφή κλπ. Θα πρέπει να το διευκρινίσουμε και καταλαβαίνετε ότι ο καθένας έχει δεν είναι απλό το πράγμα. Το είδαμε κατά τη διάρκεια της για τη, διάρκεια, για τη δικαιώματα των καταναλωτών. Ε, αλλά είναι απαραίτητο ακριβώς όχι μόνο για να υπάρξει μια εμπιστοσύνη, αλλά για να μπορέσουμε να έχουμε νέες παρόμοιες ε, επιχειρήσεις ε, γιατί το Amazon όπως ας πούμε που είναι στην πρωτοπορία μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα αλλά για ένα μικρό οργανισμό, μια μικρή εταιρεία, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και αυτό τους περιορίζει σχετικά με την ανταγωνιστική τους φύση. Και ακόμα ένα κέντρο ε, επαφής, ε, η θηρίδα Solvit και να είναι και ο σε περίπτωση προβλήματος. Ε, δεν έχουμε μόνο μονοπόλιο τώρα πια που απλά και μόνο έπρεπε να πάει κανείς στα ταχυδρομεία του. Τώρα υπάρχουν διάφοροι που επεμβαίνουν και οι οποίοι είναι υπεργολάβοι ουσιαστικά και μάλιστα πολύ συχνά είναι υπεργολάβοι και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτή τη διάσταση τη διαμεθοριακή. Ολοκλήρωσα. Λοιπόν, για τις τεχνικότερες λεπτομέρειες τώρα θα πρέπει να έχουμε ένα, μια τυποποίηση ευρωπαϊκή ώστε να μπορούν να συνεργαστούν όλα να υπάρξουν, ε, να πούμε τυποποίηση ποιοτική και μια πραγματική ανεχνευσιμότητα όσον αφορά την παράδοση αυτών των δεμάτων. Κάτι που δεν θα πρέπει να παραλείπουμε είναι και η κοινωνική πτυχή, γιατί εκεί γίνονται πάρα πολλές ε, παραβιάσεις όσον αφορά το ε, δικαίωμα εργασίας γιατί υπάρχουν ε, αρνητικές συνθήκες εργασίας με μη κατάλληλο καθεστώς εργαζόμενου και αυτό δεν είναι και υπέρ της καλής ποιότητας της υπηρεσίας γι' αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό το πράγμα ώστε να μην παροτρύνουμε για παρόμοιες μη θετικές ενέργειες και να υπάρξει μια κατάλληλη συνεργασία. Αυτά και σας ευχαριστώ. <laughs> Ευχαριστώ. Θα είμαι σχετικά σύντομη, διότι ήδη πολλά είπαν. Πρόκειται για νέα αγορά και πρέπει να φροντίσουμε και την ενημέρωση των καταναλωτών και βεβαίως και τις ανάγκες των εμπόρων που δραστηριοποιούνται μέσω του διαδικτύου αλλά και των μεταφορέων. Εξήγησαν πολλά ήδη οι προλαλήσαντες και οι προλαλήσαντες. Ε, πολύ ευχαρίστως θα συνεχίσω τη συνεργασία και για την ώρα αρκούμε σε αυτά, άλλωστε πρέπει να φύγω να πάω σε άλλη συνεδρίαση. Εσείς κύριε Κράμερ, αν μπορούμε να είμαστε σύντομοι τόσο το καλύτερο. Η σκιώδη συγγήτρια Λίχτενμπέργκερ είναι στην άλλη επιτροπή και, και με παρακάλεσε να την εκπροσωπήσω. Η αγορά αυτή χαρακτηρίζεται από προβλήματα μεταξύ άλλων στις διαμεθοριακές μεταφορές. Για παράδειγμα, η DHL προβαίνει σε διάκριση ανάμεσα στα κερδοφόρα τμήματα της αγοράς και στα λιγότερο κερδοφόρα τμήματα της αγοράς. Ουδόλως ενδιαφέρεται να παραδίδει για παράδειγμα σε νησιωτικές περιοχές. Γι' αυτό και πρέπει να το τονίσουμε και να ε, τονίσουμε που εντοπίζονται τα σφάλματα, οι ελλείψεις και να φροντίσουμε να είναι ίσες οι όροι ανταγωνισμού. Άλλωστε είναι γνωστό ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο ίντερνετ και φοροδιαφεύγουν ή τουλάχιστον φόρο αποφεύγουν και παραβιάζουν σημαντικές διατάξεις της αγοράς εργασίας. Τα έσοδά τους τα μετακινούν σε φορολογικούς παραδείσους. Εκεί όπου αποκομίζουν τα κέρδη τους δεν καταβάλουν φόρους. Μπορώ να σας πω και ονόματα. Emerson, Starbucks. Διότι προσφέρουν φτηνές τιμές αλλά σε βάρος των εργαζόμενων. Ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας ε, υπασχολήσει εδώ βεβαίως είναι και η προστασία του κλίματος και η ανάγκη μείωσης των εκπομπών αερίων. Υπάρχουν εφόσον το επιθυμούμε και καλύτερες λύσεις για τη μεταφορά. Είναι αυτά τα post-box τα οποία, ε, ε, όπου μπορεί κανείς να πάει και να παραλάβει το πακέτο του ανά οποιαδήποτε ώρα. Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας. Υπάρχουν λοιπόν και άλλες ε, τεχνολογίες. Όλοι σήμερα λίγο πολύ έχουν ε, κινητά τηλέφωνα. Όταν λάβω την πληροφορία ότι ήρθε το πακέτο μου και βρίσκεται στο τάδε μέρος, μπορώ να πάω να το πάρω. Αυτό και εμένα με εξυπηρετεί και μάλιστα μπορεί να μείνει εκεί ας πούμε μια ολόκληρη εβδομάδα ώστε να πάω όταν με βολεύει. Προς αυτή την κατεύθυνση θεωρούμε ότι πρέπει να κινηθούμε. Ζέλερ. Ζήλε μάλλον. Εμείς νομίζουμε ότι καλά λειτουργεί η αγορά αυτή. Είναι πολύ ανταγωνιστική. Υπάρχει ευρύ φάσμα παρόχων υπηρεσιών και αυξάνεται πολύ το λιανικό εμπόριο στο διαδίκτυο. Οποιαδήποτε νομοθεσία ενδέχεται να έχει αντικές επιπτώσεις και να είναι αντικίνητρο για οποιαδήποτε εξέλιξη. Εμείς νομίζουμε ότι καλώς αντιδρούν στις πιέσεις των καταναλωτών και αναπτύσσουν νέες υπηρεσίες. Η Κομισιόν έχει προβλέψει ορισμένες οδηγίες στην Πράσινη Βίβλο που αντιμετωπίζουν και τους φραγμούς στο ηλεκτρονικό εμπόριο, κάτι το οποίο εφόσον καταργηθούν δηλαδή αυτά θα ωφελήσουν τους καταναλωτές και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Εμείς λοιπόν είμαστε ικανοποιημένοι με την αγορά αυτή. Βέβαια είμαστε και ανοιχτοί σε οποιαδήποτε μορφής συνεργασία. Δεν έχω άλλους εγγεγραμμένους ή άλλες εγγεγραμμένες. Κομισιόν, ναι, όχι, όχι, ωραία. Και Νταντά. Χρονοδιάγραμμα. Σχέδιο εκθέσεως 5 Σεπτεμβρίου. Κατάθεση τροπολογιών έως 18 Οκτωβρίου. Ψηφοφορία 5 Νοεμβρίου. Στην Επιτροπή δηλαδή. Αν σας ικανοποιεί το χρονοδιάγραμμα, προχωρούμε έτσι. Ωραία λοιπόν. Ωραία, μου εξοικονομήσατε κάποιο χρόνο. Προχωρούμε στο δεύτερο μέρος των σιδηροδρόμων. Ανταλλαγή απόψεων. Μήπω μπορεί κάποιο να ψάξει να βρει του διάφορους εισηγητές, Ιδίω Αλκαντράουι και Γκρόσου θα μας βοηθήσει πολύ. Could I ask the, Mrs. Wills, do you know if Mr. Κυρία Βίλς, γνωρίζετε αν θα έρθει ο κύριος Κόλιτσεκ. Δεν θα έρθει, θα μιλήσω εγώ για λογαριασμό του. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε με τον ίδιο τρόπο, όπως και χθες. Έξι λεπτά για τους εισηγητές, τέσσερα λεπτά για κάθε έναν από τους σκιώδες εισηγητές και μετά δύο λεπτά για κάθε ένα από τα μέλη της Επιτροπής που θα θέλει να παρέμβει και τέλος ο εκπρόσωπος της Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έχει το λόγο να μας κάνει μια γενικότερη επισκόπηση. Επρόκειτο να ξεκινήσω με το PSO, την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, αλλά θα ξεκινήσω με τη διαχείριση και το άνοιγμα της αγοράς για τη μεταφορά, την εγχώρια σε εθνικό επίπεδο των επιβατών. Παρακαλώ, κύριε Αλκεσίλη, έχετε το λόγο. Ναι, χαίρομαι που οργανώθηκε αυτή η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για ένα θέμα που θα μπορούσε να επηρεάσει τα πράγματα ιδιαίτερα για εκατομμύρια ταξιδιώτες ακριβώς τη στιγμή εκείνη που μετακινούνται. Εμείς, η κοινή στόχη μας θα πρέπει να είναι να βοηθήσουμε ώστε να ενισχυθούν οι σιδηρόδρομοι στις, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι να αποδυναμωθούν και για την οργάνωση της εθνικής μεταφοράς. Δεν είναι αυτός σκοπός. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι πρώτες ε, εμπειρίες δεν ήταν πάντα θετικέ Αυτό το δίκτυο, η οργάνωσή τους, ε, ε, για το άνοιγμά τους, τη φιλαδροποίησή τους, όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να επηρεαστούν ανάλογα σε κάθε μέλο. μέλος. Υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία εδώ και 20 χρόνια πειραματίζονται με τον ανταγωνισμό αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες στις οποίες αποτελεί μονοπόλιο ακόμα σε υδρόδρομος. Ιδεολογική τοποθέτηση λοιπόν που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγχυση αλλά χρειάζονται οικονομικές προσπάθειες για αποτελεσματικότητα και ποιότητα. Και κάτι τέτοιο θα μπορούσε βέβαια να ποικίλει από τη μία χώρα στην άλλη. Πάντως θεωρώ ότι χρειάζεται να έχουμε παροτρύνσεις και μια ρεαλιστική αντιμετώπιση και ειδικότερα για ό,τι αφορά τις ε, συμφωνίες με το δημόσιο που δεν θα πρέπει να έχουν να κάνουν απλά και μόνο με μια ανοιχτή πρόσβαση σχέση και θα ήθελα να μιλήσω για μερισμένα πράγματα για το άνοιγμα της αγοράς, κυρίως στις περιοχές εκείνες που δεν έχουν να κάνουν με τα κανονικά, με τις κανονικές συμβάσεις, τις κανονικές συμφωνίες. Θα πρέπει να έχουμε το open access, ε, την ελεύθερη ανοιχτή πρόσβαση, αλλά Ταυτόχρονα τα κράτη-μέλη εκεί που δεν είναι δυνατό κάτι τέτοιο πρέπει να υπάρχουν επιλογές και αυτό υπάρχει στη Γερμανία. Τα κράτη-μέλη ε, επιλέγουν μια δυνατότητα ανοιχτής πρόσβασης που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε περιοχές που συμβάλλονται με μια κατάλληλη συμφωνία και να υπάρξει και μια οικονομική ισορροπία και να μην υπάρχουν κίνδυνο ε, για ορισμένα συμφέροντα. Εδώ και στην πρόταση της Επιτροπής αναφέρεται άλλωστε ότι εάν κάποιος νέος που μπαίνει στην αγορά και θέλει να χρησιμοποιήσει το δίκτυο, τότε χρειάζεται μια επαλήθευση, ένας έλεγχος εάν κινδυνεύουν οικονομικά συμφέροντα και αν χρειάζεται ένας περιορισμός. Μία τρίτη δυνατότητα που δεν προβλέπεται αλλά είναι σημαντική, ε, ένα κρατος θα πρέπει προκαταρτικά να αποφασίζει ότι εκείνος ο οποίος ε, είναι συμβαλόμενος ε, θα μπορεί ή όχι να κάνει χρήση ενός μονοπολίου ουσιαστικά για μια ορισμένη όμως περίοδο της συμφωνίας του και για μια ισορροπία οικονομική. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται και όχι μόνο με εκτελεστικές πράξεις. Όσον αφορά την οργάνωση τώρα των σιδηροδρόμων θα ήθελα να αναφερθώ στη διατήρηση σημαντικών αρχών όπως τη δυνατότητα ε, επιδοτήσεων, ενισχύσεων κλπ. Πολλαπλών μάλιστα να δούμε και τι γίνεται, πώς μπορεί κανείς να ενισχύσει την όλη προσπάθεια και εκ των προτέρων με εκ των προσπάθειες και βέβαια το κεφάλαιο αυτό είναι ακόμα ανοιχτό αλλά θα πρέπει νομίζω να επιδηθεί ο κατάλληλος ρεαλισμός σχετικά με τις υπηρεσίες που θα πρέπει να προστατεύονται ποιες ναι, ποιες όχι και αν όσοι εργάζονται μπορούν να μεταπηδούν σε άλλη εταιρεία εάν το επιθυμούν. Χρειάζεται όμως μια κάποια αυτονομία, θα πρέπει να εξετάσουμε κανονικά όπως πρέπει τους κανόνες του παιχνιδιού. Ίσως ε, χρειάζονται και εξαιρέσεις όπως τα πράγματα όταν αφορούν τις μικρές τοπικές επιχειρήσεις οι οποίες εργάζονται ακριβώς και συνεργάζονται σε αστυνομικά θέματα. Διαφορετικά θα μπορούσαν να δαπανούν πολλά χρήματα και να μην έχουν κάτι το θετικό. Και ακόμα την κοινωνική πτυχή που προβλέπεται η δυνατότητα από τα κράτη-μέλη να ενεργήσουν όπως πρέπει ώστε να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις και να σέβονται ορισμένες ελάχιστες ε, προδιαγραφές για να υπάρχουν και ίσοι όροι και ευκαιρίες. Ακριβώς δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε, να παρακάμπτουμε την κοινωνική πτυχή. Χρειάζονται και προσπάθειες κατάλληλες προς την κατεύθυνση αυτή. Ακόμα θεωρώ ότι απαιτείται να λυθούν θέματα που έχουν να κάνουν με τους επιβάτες και με την πρόταση της Επιτροπής για την διαμεθοριακή συνεργασία, όπως παραδείγματος το δίκτυο των διαχειριστών της όλης οργάνωσης και των ρυθμιστών. Είναι μια θετική ιδέα, συμφωνώ. Υπάρχουν όμως και πρακτικής φύσεως θέματα τα οποία χρειάζεται να επανεξεταστούν όσον αφορά τις λεπτομέρειες τους. Αυτά θέλω να πω εισαγωγικά και με το σκέτο συγητή μπόρεσα να συνομιλήσω και ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλό για αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάντσεν για το ΕΡΚ. Τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο στόχος της τέταρτης συνδρομικής δέσμης είναι να πετύχουμε την ενιαία σιδηροδρομική αγορά. Ελπίζουμε να είναι και η τελευταία. Για το στόχο αυτό μπορούμε να συνεργαστούμε και ανάμεσα στους stakeholders να δώσουμε απαντήσεις και οι πολίτες πρώτα απ' όλους μέσω μια κατάλληλη βελτίωσης των υπηρεσιών χωρί να αυξηθούν όμω οι τιμέ και διάφορε εταιρείε με όλε αυτέ τι προδιαγραφέ και την όλη διαδικασία χαμηλό κόστο για όλα αυτές τι προμήθειες ανάμεσα στους προμηθευτές και πελάτε και τα κράτη-μέλη και να μην ρίξουν το βάρο στον εθνικό προπολογισμό, στον δημόσιο προπολογισμό και σχετικά με το άνοιγμα τη εθνική μεταφορά ακριβώ και για την governance αυτή τη όλη υποδομή. Χρειάζεται όλα αυτά να συμμετάσχουν πρέπει και με κατάλληλα μέτρα ακριβώς σε σχέση με τους στόχους και να μπορούν να υποστηριχθούν, μπορούν να, ε, μπορούμε να τους ε, αναλάβουμε ε, από οικονομικής πλευράς. Και τώρα το άνοιγμα της αγοράς. Εκεί θα πρέπει να πετύχουμε μια συμφωνία για τις εθνικές μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών. Όσο γίνεται πιο πλατιά συμφωνία και για τις και για τη συμβατική αλλά μακράς απόστασης μεταφορά σύντομα, όπως πρέπει, καθορισμένα και όχι πέρα από το 2019. Άρα λοιπόν θετικό θεωρώ ότι δεν υπάρχει πια διάκριση ανάμεσα σε εθνική και σε διεθνή υπηρεσία μεταφοράς επιβατών. Μια ρήτρα όμως αμοιβαιότητας θα πρέπει να προβλεφθεί στη μεταβατική περίοδο γιατί οι εθνικές νομοθεσίες δεν έχουν ένα χαρακτήρα σε αυτό και θα πρέπει αυτή η ρήτρα να περιλαμβάνει και άλλα σημεία αυτή η αμοιβαιότητα και προς χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι ακόμα δεύτερο, μια, ε, το PSO, μια κατάλληλη ισορροπία για να έχουμε την κατάλληλη εγγύηση ανάμεσα στο δίκτυο αυτό και στις ε, δημόσιες ε, με το δημόσιο. Πρόκειται για κάτι λεπτό, ευαίσθητο. Χρειάζεται να το εξετάσουμε λεπτομεριακά, να το συζητήσουμε, να λάβουμε υπόψη μας τον ειδικό χαρακτήρα σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό το governance, τη διαχείριση ακριβώς ε, για τον διαχειριστή. Ε, πρέπει να δούμε τα όσα έχουν εισαχθεί, τα έχουν, έχουν ισχύσει και θα πρέπει να δούμε πόσο αποδεσματικά όλα αυτά, πόσο μπορούν να γίνουν ανεκτά οικονομικά. Κάτι που δεν κατάλαβα ακόμα για πόσους μέχρι τώρα ακούσαμε εδώ και θα πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειες. Εάν υπάρχουν ελλακτικέ λύσεις θα πρέπει όλα αυτά να τα εξετάσουμε λεπτομεριακά ώστε στο τομέα και οι χρήστες και οι φορολογούμενοι να μην υποστούν το βάρος μιας μεταρρύθμισης και μετά δεν υπάρχει ίσως και τόση καλή ποιότητα το impact assessment, impact assessment ε, της Επιτροπής. Ε, θα πρέπει να δούμε πώς ορισμένες ρυθμίσεις μπορούν να ενισχυθούν σύμφωνα με το RECAST ε, πάνω απ' όλα του ρυθμιστή και θα πρέπει να ενισχύσουμε όλα αυτά που γίνονται σε εθνικό επίπεδο, να είναι ανεξάρτητα και ένας Ευρωπαίος ισχυρός ρυθμιστής που να μπορεί να βάλει τελικές αποφάσεις την περίπτωση που υπάρχουν αντιπαραθέσεις και σε εθνικό επίπεδο. Εδώ κάτι ακόμα είναι να υπάρξουν οι βασικές λειτουργίες να διατηρηθούν ε, όπως να δούμε ακριβώς ε, την πορεία και τα διόδια που θα πρέπει όλα αυτά να διαχειριστούμε διάφανα από όλους, για όλους και κυρίως απέναντι στον ρυθμιστή. Τέσσερα λεπτά εξ ονόματος των φιλελεύθερων, ο κύριος Τομόλσοφ. Τρεμόσα ή Μπαλσέλ. Ευχαριστώ. Μιλώ εξ ονόματος του κυρίου Φίλιπ Ντεμπάκερ. Δεν συμμερίζομαι 100% της απόψεις του για την ε, διαχείριση και διακυβέρνηση, αλλά θα ήθελα να διαβάσω ε, τις σημειώσεις που μου έδωσε. Θέλει λοιπόν να ευχαριστήσει τον εισηγητή καταρχάς και για τη δουλειά του αλλά και για τις συναντήσεις που είχατε εσείς κύριε εισηγητά μαζί του. Θεωρεί ο Φίλιπ Τεμπέικερ ότι το τέταρτο, η τέταρτη σιδηροδρομική δέσμη είναι εξαιρετικά σημαντική. Θεωρεί επίσης ότι συμφωνούμε όλοι ότι χρειάζεται να ανοίξει η αγορά αυτή και το ερώτημα είναι το πώς. Σίγουρα όμως όλοι συμφωνούμε για τα ωφέλη του ανοίγματο της αγοράς μετά τη μεταφορά τη διεθνή των επιβατών και μετά τη μεταφορά των εμπορευμάτων, δύο κλάδοι οι οποίοι θεωρητικά έχουν ανοίξει, το επόμενο σωστό και καλό βήμα είναι το άνοιγμα της αγοράς της υδροδρομικής και σε αυτό συμφωνούμε. Το θέμα είναι το πώς και άρα θα πρέπει να βρεθεί συμφωνία για την έκθεση αυτή. Ο Φίλιπ Τεμπέικερ επίσης καλωσορίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει όμως την εξή ανησυχία και ίσως είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να μοιραστώ μαζί σας. Θεωρεί ότι ενδεχομένως ορισμένα κράτη-μέλη μπορεί να μπουν στον πειρασμό να χρησιμοποιήσουν τον κανονισμό για τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, το Public Service Obligation, για να μπλοκάρουν την είσοδο νέων φορέων εκμετάλλευσης στην αγορά. Ότι ίσως ο κανονισμός δηλαδή για το PSO χρησιμοποιηθεί από ορισμένα κρατημέλη για να υψωθεί ένα εμπόδιο και να μην μπορούν οι νέες εταιρείες να μπουν στην αγορά. Ως προς τη διαχείριση, η πλήρη κάθετη, ε, ο πλήρης, ε, κάθετος διαχωρισμός είναι το καλύτερο για να έχουμε ένα παιχνίδι επίσης όρης για όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους. Θεωρεί ο Φίλιπ Ντεμπέκερ ότι αυτό από πολιτική σκοπιά δεν είναι εφικτό. Επομένως, στηρίζει την πρόταση την, ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, θέσπιση ισχυρών προϋποθέσεων και προδιαγραφών. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και προς την ε, μεγαλύτερη χρηματοοικονομική διαφάνεια ως προς τις χρηματοδοτικές ροές, παρόλο που πάλι δεν θα αποφευθεί η διασταυρούμενη, αν επιδότηση συμφωνεί με την πρόταση επέκτασης των αρμοδιοτήτων ε, και την αύξηση της ανεξαρτησίας των μάνατζερ υποδομών, κάτι το οποίο δεν, των διαχειριστών δηλαδή υποδομής, το οποίο δεν είναι προφανές σε όλη την Ευρώπη, είναι κάτι που μόλις τώρα ξεκινάει στις χώρες του Νότου και για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς είναι απαραίτητη η ανεξαρτησία και η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των διαχειριστών υποδομών. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των σιδηροδρομικών της σιδηροδρομικής αγοράς. Αυτές είναι οι απόψεις του κυρίου Ντεμπέικερ. Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέψετε θα προσθέσω και τη δική μου προσωπική άποψη από εδώ και στο εξή για να μην ξαναπάρω το λόγο αργότερα. Όπως θα γνωρίζετε, αγαπητοί συνάδελφοι, ζήτησα τη σύσταση ενός φορέα ευρωπαϊκού ρυθμιστικού για τα των σιδηροδρόμων. Δεν ε, εκφράζω την άποψη του Φίλιπ Τεμπέκερ, εκφράζω τη δική μου άποψη. Αυτό έχει, γίνει, ε, έχει ήδη υποθέσει στη συζήτηση επί αναδιατύπωση πριν από τρία χρόνια. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο λοιπόν να έχουμε ένα ευρωπαϊκό ε, ρυθμιστικό φορέα, μια ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή. Ευχαριστούμε εξ ονόματο των Πρασίνων η κυρία Ντουράν για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε για την, ε, σεβασμό αυτό η Επιτροπή στην πρότασή της ε, λέει ότι είναι αξίωμα ότι ο ανταγωνισμός είναι κάτω παραδοητικό εξορισμού και μας προτείνει όπως και το εξήγησε ο εισηγητής μας τρόπο το πώ θα κατακαιρματιστεί αυτή η υπηρεσία που κατά την άποψή μου είναι κάτι αντιπαραγωγικό. Το όφελο που θα περίμενε κανείς, που περιμένει η Επιτροπή από τον ανταγωνισμό, δεν είναι σίγουρο αυτό το πράγμα ότι θα αντισταθμίσει κάθε πρόβλημα και υπερβολικό κόστος λόγω της κατάτμισης αυτή των υπηρεσιών ε, κατά την προκήρυξη διαγωνισμών και άλλα παρόμοια. Θα πρέπει να δούμε πού γίνονται όλα αυτά τα πράγματα και σε ορισμένε χώρες. Ε, δεν έχουμε μόνο μεγάλες χώρες στην Ευρώπη, έχουμε και μικρές χώρες. Ιδιαίτερες διαφορές και σε ορισμένε χώρες θα έχουμε μια τρομερή κατάτμιση σε αυτούς του προκήρυξης διαγωνισμών και που θα διαλύσουν το σύστημα κομματάκια-κομματάκια και θα είναι αρνητικό αυτό αυτό το δίκτυο να το κάνουμε κομμάτια-κομμάτια εκεί που είναι δύσκολο να έχουμε έναν συντονισμό ανάμεσα στους διαχειριστές αυτών και στις εταιρείε δρομόνων και να τους επιβάλλουμε επίσης ε, να έχουμε διαφορετικά τμήματα είναι κάτι το πολύ δύσκολο και ακόμα η κοινωνική πτυχή αυτό σε περίπτωση προκύψη διαχωρισμού το ποιος θα αναλάβει το σύστημα να δούμε αυτό το υλικό είναι πολύ δεσμευτικό το κείμενο θα πρέπει αυτές οι επιχειρήσεις, αυτές οι εταιρείε να το πάρουν αυτό το υλικό ως έχει. Ενώ έχουμε κοινωνικά μέτρα τα οποία α, αυτά είναι προαιρετικά. Εδώ δεν ε, είναι κάτι το συνεκτικό και θα πρέπει ε, σε αυτό αυτόματα ότι συμπεριλαμβάνεται και για την κοινωνική πτυχή. Λέμε ό,τι θέλετε κάνετε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, όσον αφορά τις υποχρεώσεις για πλευρά δημοσίου, αυτό το πρότυπο που θέλουν να μας επιβάλλουν έτσι εννέα σε όλους είναι κάτι επικίνδυνο, ούτε την, ε, δεν, δεν σέβεται τίποτα ε, και θα πρέπει να δούμε την εργασία που γίνεται πάνω σε αυτό για τους δρόμους ώστε να μπορέσουμε να τα όλα αυτά τα πράγματα για να μπορούμε να σεβαστούμε, να μην υπάρξει μια κατάτμιση αυτής της υπηρεσίας σε πολύ μικρά μέρη και που θα προκαλέσει υπερβολικό κόστος και δυσκολίες συντονισμού παρά θετικά στοιχεία και ωφέλη όσον αφορά αυτές τις γραμμές ε, στις υπηρεσίες υδροδρόμων. Ο κύριος Βλάσσερ από τους Ιδετικούς, ο Ρόμπερτ, εσύ τον εκπροσωπείς φαντάζομαι, έτσι δεν είναι. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι ένας πυλώνας που γνωρίζω πάρα πολύ καλά, γνωρίζω πιο πολύ τα τεχνικά θέματα. Ωστόσο, για τη μεταφορά των επιβατών έχω κάποιες ερωτήσεις και κάποια σχόλια να κάνω θα έπρεπε να έχουμε υπόψη μας ότι το γεγονός το εξής. Διαφέρει η κατάσταση των επιβατών ανά την Ευρώπη, σε πάρα πολύ μάλιστα. Σε ορισμένες χώρες κανείς δεν ενδιαφέρεται για τη μεταφορά των επιβατών και χωρίς επιδοτήσεις γραμμών οι χώρες αυτές δεν θα καταφέρουν ποτέ να εξυπνήσουν τον ενδιαφέρον των εταιριών για να μεταφέρουν επιβάτες στο εσωτερικό της επικράτειάς τους. Υπάρχουν αγορές πολύ ενδιαφέρουσες όπως είναι η Benelux, η Γερμανία, η Γαλλία, αλλά η κατάσταση είναι διαφορετική αλλού. Δεν είναι όλα όπως εδώ και θα πρέπει ε, να γνωρίζουμε ότι ένας κανονισμός για το PSO, για την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας θα μπορούσε να συνεπάγεται τον περιορισμό της πρόσβασης στην αγορά σε κάποιες άλλες αγορές. Να είμαστε λοιπόν εξαιρετικά προσεκτικοί παρακαλώ. Από εκεί και πέρα, πόσο μακριά πρέπει να φτάσουμε με τον κατακαιρματισμό. Ίσως τον πρώτο λόγο θα πρέπει να έχουν οι ίδιοι επιβάτες, οι χρήστες της ε, σιδηροδρομικής υπηρεσίας. Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται οι ανταποκρίσεις μεταξύ περιφερειακών τρένων και εθνικών τρένων. Οι επιβάτες θα πρέπει να αποφασίσουν γι' αυτά, να έχουν τον πρώτο λόγο. Κατά τη γνώμη μου το ελβετικό σύστημα είναι εξαιρετικά καλό, έχει πολύ καλό δίκτυο μεταξύ των μεγάλων πόλεων και των διεθνών συνδέσεων από τη μία και των περιφερειακών συνδέσεων εδώ, εντός της χώρας από την άλλη. Εάν κρατήσουμε κι εμείς αυτό το πνεύμα, τότε θα κάνουμε πολύ καλή δουλειά. Ο δρόμος είναι μακρύς μπροστά μας για να φτάσουμε στο τέλος. Εύχομαι επιτυχία στον εισηγητή. Κυρία Ζήλερ και κυρία Βίλτς, τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ. Συνεχίζει η Κομισιόν την προσπάθεια απελευθέρωσης στον τομέα των σιδηροδρόμων. Ανοίγει λοιπόν ένα ακόμη κεφάλαιο σε αυτή την χωρίς συμβιβασμούς πολιτική που ακολουθεί την ενδιαφέρει βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών υπέρ των επιβατών, την ενδιαφέρει να λάβουν περισσότερες δουλειές οι ιδιωτικές επιχειρήσεις σε βάρος των δημόσιων επιχειρήσεων σιδηροδρόμων, των οποίων τους αφαιρείται ούτως ή άλλως και κάθε περιθώριο ελιγμών. Είμαι πεπισμένη, ένα λεπτό, ότι με αυτή την πρόταση της Κομισιόν η προσπάθεια που γίνεται είναι να συνεχιστεί η προσπάθεια που άρχισε με την αναδιατύπωση της οδηγίας περισσυδροδρόμων του Δεκεμβρίου 2012. Βλέπουμε αυτό το unbundling και την ε, νομική διάκριση μεταξύ management και ε, λειτουργίας του σιδηροδρόμου. Εκεί ούτως ή άλλως είχε καταλήξει η ομάδα μου στην ε, απόρριψη του συμβασμού γιατί δεν περιλάμβανε τα στοιχεία που ε, θέλαμε να δούμε. Ο μέχρι τώρα απολογισμός της προσπάθειας αυτής απελευθέρωσης δεν ε, θεωρούμε ότι επιτρέπει να προχωρήσουμε στην υιοθέτηση του μοντέλου της απόλυτης διάκρισης μεταξύ δικτύου και διαχείρισής του. Για μας, ως Ενωτική Αριστερά NGL, ήταν πάντα καθαρό ότι ο σιδηρόδρομος είναι ένα ενιαίο σύνολο που δεν μπορεί να χωριστεί σε κερδοφόρα και μη κερδοφόρα τμήματα. Μόνο μέσα στα πλαίσια μιας δημοκρατικά ελεγμένης πολιτικής μεταφορών μπορούμε να διασφαλίσουμε το μέλλον των μεταφορών. Unternehmen die Möglichkeit von και που βαίνει και το θέμα των εργαζόμενων. Πού θα πάνε οι εργαζόμενοι όταν θα διαλυθούν οι δημόσιες επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό και δεν μπορεί να μείνει ανεπίλητο, διότι η δυνατότητα απασχόλησης ορισμένων εργαζόμενων μάλλον εξατμίζεται, κάτι το οποίο σημαίνει την απώλεια ε, προσοντούχων και εμπειρών συνεργατών. Τέλος, έρχομαι σε μια δήλωση του Επιτρόπου Κάλας σχετικά με τη δημιουργία ενιαίου σιδηροδομικού χώρου και ανοίγματο της αγοράς για τις εσωτερικές μεταφορές σιδηροδρόμων, εμπορευμάτων και προσώπων. Δεν φοβείται ότι θα επιδεινωθούν οι συνθήκες εργασίας. Ωστόσο, οι εμπειρίες των χωρών μελών που άνοιξαν τις σιδηροδρομικές αγορές τους έδειξαν ότι αυτό οδήγησε, λέει στην ανακοίνωση τύπου του ο Επίτροπος, ότι υπήρξε βελτίωση. Αυτό, ωστόσο, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας, δεν είναι ορθό, διότι έδειξε εκεί ότι ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός επιφέρει ζημία, διότι μειώνεται το επίπεδο ασφάλειας προκαλείται κοινωνικό dumping και dumping μισθών και δεν εξυπηρετούνται παρά μόνο οι επικερδείς διαδρομές. Εγώ εξακολουθώ και είμαι αντίθετη με οποιαδήποτε τέτοια πολιτική. Κύριε Πρόεδρε, συναδελφοί, η γερμανική και η γαλλική τοποθέτηση. Εδώ δεν προβλέπεται μια ε, απομάκρυση ανάμεσα στο διαχειριστή και εκείνους που ασχολούνται με τις μεταφορές. Και στην αρχή ήταν μια διάμεση φάση για να υπάρξει αυτή η κατομμυσή. Ενώ είναι τελευταία φάση, ε, είναι τελευταία φάση. και τα holdings ε, διατηρούνται και για ορισμένους που διαχειρίζονται αυτά με την ξεχώρισμα του κόστους ανάμεσα σε εκείνους που ασχολούνται στην ίδια ομάδα όμως. Και θεσμική αυτή απομάκρυση θα είναι η βασική αρχή, αλλά όλα αυτά θα μπορούσαν να συνεχίσουν να υπάρχουν αν υπάρχουν ρήτρες διαφύλαξης αυστηρές για μια ανεξαρτησία οικονομική, νομική, επιχειρησιακή σε αυτή την δομή. Και οι συζητήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ξεκινάει όμως, όπως το κάνει τώρα, την εξέταση στο του σχετικού κειμένου. Θεωρώ ότι αυτός ο τελικός στόχος που είναι αυτή η διαχείριση ανάμεσα και την εκμετάλλευση δεν είναι σύμφωνα με αυτά που μας απασχολούν οικονομικά και κοινωνικά που έχουν να κάνουν με υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος που θέλουμε αύριο να προτείνουμε στην Ευρώπη. αλλά με υπόψη μας αυτές τις εμπειρίες που είχαμε σε διάφορες χώρες που νομίζω ότι ήταν αρνητικές κατά την απόψή μου. Αυτός ο διαχωρισμός ε, ε μας δημιουργήσει περισσότερο πολύπληκες καταστάσεις στη διαδικασία. Ε, θα γίνει κάπως άκαμπτο το όλο θέμα επειδή θα υπάρχει κατάλληλη συνεργασία και ανάλογη ανάληψη. Εδώ δεν θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν περισσότερο ευαίσθητα επειδή θα υπάρχουν πάρα πολλοί που θα παρεβαίνουν και μια δομή ε, πολύ διασπασμένη. Εδώ αυτές οι υπηρεσίες δημόσιου ε, ενδιαφέροντος έχουν να κάνουν και με την όλη διαχείριση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κ. Μπαχ. Κάτι για την διαχείριση. Με απογοητεύει η πρόταση της Κομισιόν. Θα ήθελα στην πρότασή της να αφήσει ανοιχτές διάφορες δυνατότητες οι επιλογές η Κομισιόν. Μέσα στην Ευρώπη έχουμε διάφορα μοντέλα, διάφοροι σιδηρόδρομοι διαφόρων χωρών μελών. Υπάρχουν σιδηρόδρομοι που λειτουργούν θαυμάσια προς απόλυτη ικανοποίηση του κοινού, που δημιουργούν καλές θέσεις απασχόλησης και μια ικανοποιημένη πελατεία. Και με το ρικά στην αναδιατύπωση δηλαδή, δεν θέλω βέβαια να επαναλάβω τα όσα συζητήθηκαν τότε, νομίζω όμως ότι με εκείνο το αναδιατυπωμένο νομοθέτημα έχουμε πλέον μια βάση που μπορούμε να αποτρέψουμε την διασταυρούμενη χρηματοδότηση και μπορούμε να ενισχύσουμε τους ρυθμιστές. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε, να εργαστούμε στη βάση του μοντέλου αυτού, να συλλέξουμε εμπειρίες, γιατί κανένα πολίτη δεν κατανοεί πως τώρα μετά από τρει-τέσσερι μήνες ερχόμαστε να ψηφίσουμε νέα νομοθεσία. Θέλω να πω ακόμη ότι η πρόταση δεν έχει οριμάσει ακόμη. Ούτως ή άλλως υπάγεται στην επικουρικότητα διότι πρόκειται για δημόσια υπηρεσία και επομένως είναι υπόθεση της χώρας μέλους. Πλείονες χώρες μέλη αυτό έχουν δηλώσει. Και όπως είπα και με την αναδιατύπωση παραμένει το θέμα σε χώρο αρμοδιότητα των χωρών μελών λόγω επικουρικότητα. Η κυρία Σενάλοβα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να λειτουργήσουν υψηλής ποιότητας σιδηροδρόμοι δηλαδή να είναι υψηλής ποιότητας σιδηροδρομικές υπηρεσίες και σε μη κερδοφόρα τμήματα των σιδηροδρόμων. Συμφωνώ με άλλους που μίλησαν πριν ότι ανταγωνισμός και κατακαιρματισμός δεν σημαίνει ότι θα πετύχουμε το στόχο μας. Θα πρέπει να εξετάσουμε καλά τον ορισμό της δημόσιας υπηρεσίας, της καθολικής δημόσιας υπηρεσίας. Τι θα πει αυτό. Πιστεύω ότι οι δημόσιες διοικήσεις που είναι υπεύθυνε για τις δημόσιες υδροδρομικές υπηρεσίες πρέπει να έχουν την αρμοδιότητα να παρεμβαίνουν στην αγορά. Αρκούμε σε αυτά. Δύο λεπτά εσείς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για το USP, για τον κανονισμό αυτό να πω δύο πράγματα. Με συγχωρείτε. Κύριε Ζουρίμπη, θα μιλήσουμε για το PSO, την υποχρέωση παραχής δημόσιας υπηρεσίας στη συνέχεια με τον κύριο Γκρός. Και Εδώ γιατί μιλάμε. Γιατί μπερδεύτηκα κύριε Πρόεδρε. Θα σας πω γιατί μιλάμε. Μιλάμε για το άναγμα της αγοράς για τον τρόπο διαχείρισης της υδροδρομικής υποδομής και για την, το άνοιγμα της αγοράς για τη μεταφορά των επιβατών. Και όταν μιλήσουμε για αυτά, μετά θα μιλήσουμε για τη δημόσια ε, υπηρεσία. Θέλετε να μιλήσετε για την έκθεση του κυρίου Καντράουι ή θέλετε να μιλήσετε για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας. Μπορώ να μιλήσω για τη διαχείριση και διοίκηση κύριε Πρόεδρε. Ναι βεβαίως. Θα ξαναξεκινήσω το ρολόι. Μπορείτε να μας πείτε για τη διαχείριση της απόψης σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για τη διαχείριση λοιπόν. Η Επιτροπή τι προσφέρει σαν ευκαιρία. Να μην οργανωθεί κανείς σαν, σε ένα ξεχωριστό πρότυπο, αλλά έχει αυτό το συνικό τείχος ε, για να αποφύγει αυτό το ολοκληρωμένο σχέδιο να προταθεί από ένα κράτος μέλος. Κύριε Πρόεδρε, κάπως να ελαφρυνθεί αυτή η θέση, να γίνει πιο ευλή στη θέση της Επιτροπής, να μην είναι δογματική προσέγγιση και αυτό το ξεχωριστό πρότυπο σε αυτό το ολοκληρωμένο να μην το αντιπαραθέσει με την ελεύθερη επιλογή των κρατών μελών γιατί από ό,τι πιστεύω έχουμε δύο στόχους μέσω αυτού του σχεδίου για την διαχείριση μια διαφάνεια να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη σχετικά με το διαχωρισμό αυτές της λειτουργίες ε, και να μην έχουμε ένα γλίστριμα προς τον διαχειριστή. Ε, αν ε, αυτά τα πράγματα ισχύσουν, δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να απαγορεύσουμε σαν κράτος μέλος να αποφασίσει πώς θα οργανωθεί με τον καταλληλότερο γι' αυτό τρόπο, ανάλογα με το τι έχει κάνει ιστορικά, τι έχει κάνει σαν επιλογές και τι πήρα διαθέτει εδώ θεωρώ ότι το ξεχωριστό μοντέλο προς το ολοκληρωμένο να την παρθέσουμε είναι ένα λάθος και η Επιτροπή που έχει εντελώ φιλελεύθερη άποψη σχετικά με αυτό το κείμενο. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αντίφαση γιατί όταν είναι κανείς φιλελεύθερος αφήνει την ελεύθερη επιλογή στα κράτη-μέλη από τη στιγμή που αυτά τα δύο που είπα γίνονται σεβαστά για φάνεια και ανεξαρτησία από τη στιγμή που τα εγγυόμεθα αυτά. Αυτά ήθελα να πω για τη διαχείριση λοιπόν. Ελπίζω να, πως, να γίνει πιο εύκαμπτη η αρχική θέση της Επιτροπής και τα κράτη-μέλη έτσι να μπορέσουν και να τα σεβαστούν αυτά αλλά ταυτόχρονα να οργανωθούν όπως το εννοούν αυτά. Ο κύριος Κράμερ για δύο λεπτά. Βέβαια, Ματιού βλέπω χαμογελάς, υπάρχουν διαφορές απόψεων και σε όλες τις πολιτικές ομάδες. Δεν συζητούμε πλέον για το αρχικό σχέδιο της Κομισιόν. Θέλει διαφάνεια των, χρηματικών, των ε, χρηματοδοτικών ροών. Τι γίνονται τα χρήματα. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα, είμαι Γερμανός, όπου με την σιδηροδομική υποδομή αποκομίζουν οι εταιρείε μεγάλα κέρδη με τα λεφτά αυτά τι γίνεται. Εξαγοράζουν, κάποιον ανταγωνιστή. Εξαγοράζουν π.χ. στις Ενωμένες Πολιτείες μια εταιρεία λεωφορείων ή επανεπενδύονται τα χρήματα στην υποδομή για να μην εγκαταλείπονται οι σιδηροδρομικοί σταθμοί, να μην εγκαταλείπονται διάφορες γραμμές. Βεβαίως δεν μιλώ εξ ονόματος της ομάδας μου, άλλωστε αυτό συμβαίνει και σε άλλες ομάδες. Εγώ είμαι όμως υπέρ της ιδέας να ρυθμιστεί ξεκάθαρα με την ομοθεσία τα χρήματα που πάνε. Στην Νορβηγία είναι ρυθμισμένο αυτό, είναι καλή ρύθμιση γιατί θεωρείται ότι είναι καθολική υπηρεσία. Γνωρίζουμε τώρα ότι πάνω από το μισό των χρημάτων που λαμβάνουν τα γερμανικά ομοσπονδιακά κριτήδια για το σέρβις δαπανώνται για σταθμούς και για οδικές προσβάσεις. Δηλαδή δεν πάνε καν στο σιδηρόδρομο. Πρέπει η κινητικότητα ωστόσο να είναι εξασφαλισμένη. Αυτό είναι θεμελιώδες δικαίωμα του καθενός, που να μπορεί δηλαδή να υποφελείται από τη δυνατότητα μετακίνησης όπου και να κατοικεί. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα στην υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας και το άνοιγμα της αγοράς για την συνδροδρομική μεταφορά επιβατών στην επικράτεια Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ακούγοντας τις παρεμβάσεις των συναδέλφων, είναι άλλωστε και δική μου άποψη ότι έχουμε μια δέσμη μπροστά μας, θα ήταν σωστό δηλαδή, έχει ενδιαφέρον αυτό και οι δύο, δέσμες, και οι δύο εκθέσεις μάλλον να συζητηθούν και μάλιστα διακομματικά. Διότι πρόκειται για σύνολο, όχι μόνο με τούτην εδώ την έκθεση, ολόκληρο το πακέτο είναι ένα σύνολο. Αλλά και με τη συζήτηση που διεξήχθη χθες Ας μην έχουμε καμιά ψευδέστηση. Αν αύριο λόγω της τεχνολογίας ενταθούν οι διαφορές μεταξύ χωρών μελών, έχουμε και τα τεντή, έχουμε και την ε, διευκόνηση συνδέοντα της Ευρώπης, θα μείνουμε τότε στη θεωρία. Πρέπει λοιπόν να πούμε, για να είμαστε δίκαιοι, ότι ε, ζητήσαμε με μεγάλη πλειοψηφία να προχωρήσει το θέμα του ανοίγματο της αγοράς και της δομής των εταιριών και πρέπει να συζητηθούν αυτά τα πράγματα. Όχι να ζητάμε κάτι και μετά να διαμαρτυρόμαστε που έγινε. Τώρα, εγώ θεωρώ ότι με το πακέτο αυτό ανοίγεται μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να δείξουμε ότι ο σιδηρόδρομος αύριο, εφόσον γίνει πραγματικά ευρωπαϊκός, και εδώ υπάρχουν κάποιες προσεγγίσεις πολύ ενδιαφέρουσες, μπορεί όντως να οδηγήσει σε ανάπτυξη και επομένως και να ωφελήσει τον πολίτη. Έχω την εντύπωση ότι ορισμένοι συνάδελφοι δεν είναι πολύ σίγουροι. Πρέπει να στηρίξω το σιδηρόδρομό μου, πρέπει να στηρίξω τους εργαζόμενους ή καλύτερα να κοιτάξω το θέμα από την οπτική σκοπιά του επιβάτη. Νομίζω πρέπει να συνδεθούν τα συμφέροντα και των δύο πλευρών. Δεν μπορεί να είναι καθήκον της Ένωσης να καταστρέψει συστήματα που λειτουργούν και που συνεργάζονται ούτε την άλλη μεριά μπορεί να εγκαταλείψει την ε, προσπάθεια εξασφάλισης ποιότητας των σιδηροδρομικών υπηρεσιών που προσφέρονται στους επιβάτες. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Τώρα η προσέγγιση στο στόχο αυτό γίνεται από διάφορες πλευρές. Για μένα σημαντικός είναι και ο ρόλος των τοπικών αρχών. Αυτές είναι που πρέπει να φτιάξουν σχέδια, να σχεδιάσουν συστήματα που να είναι και πολυτροπικά. Ε, να έχουν δηλαδή σαν πυρήνα τη συνεργασία των διαφόρων τρόπων μεταφορών. Ο δε πολίτης, ή μάλλον η, ε, η, τοπική αρχή να είναι σε άμεση επαφή με τον πολίτη. Ο πολίτης να πει του αρέσει αυτό που προτείνει η αρχή ή όχι. Αυτό πρέπει να γίνει. Το ίδιο και, και για τους κανόνες, για, για τα επίπεδα Τη ποιότητα, όπου πρέπει να μπουν όλα, δηλαδή και οι περιβαλλοντικοί κανόνες και ούτω καθεξής. Εμεί δεν θέλουμε να μειωθούν αυτά. Το δεύτερο που είναι σημαντικό είναι η κατανομή. Όπως και άλλοι συνάδελφοι, εγώ ζητώ πολύ μεγαλύτερη ευελιξία. τα προτινόμενα εδώ δεν είναι καλά ούτε για τις μικρές ούτε για τις πολύ μεγάλες χώρες. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες των διαφόρων χωρών μελών. ο χώρος που προσφέρεται, αυτό το bassin de vie όπως λένε στα γαλλικά, δεν μπορεί να καθοριστεί μέσα από πολιτικές δομές. Πρέπει να είναι πολύ καλύτερα προσαρμοσμένο στην καθημερινή πραγματικότητα. Τρίτο, πρέπει να δικαιολογείται και η χρηματοδότηση για τις υπηρεσίες αυτές. Εδώ εντοπίζεται η μεγάλη ευθύνη της πολιτικής και των τοπικών αρχών. Ποιότητα, βελτίωση της ποιότητας η χρήση που επιφυλάσσουν στα χρήματα των φορολογουμένων, που πρέπει να καταλήγουν στους επιβάτες, και όμως απέναντι στους φορολογούμενους. Αυτό που προτείνω εγώ ως μεθοδολογία είναι ευνοϊκό, είναι δηλαδή φθηνό και εδώ νομίζω ότι είναι σωστή η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εφόσον δεν είμαστε δογματικοί. Έρχομαι τώρα και στην άλλη έκθεση επιθυμώ να διεξαχθεί συζήτηση για την αποτελεσματικότητα, όχι οχυρωμένη δογματικά, και σε ό,τι αφορά την δομή και σε ό,τι αφορά την ανάθεση των υπηρεσιών. Θα φτιάξουμε τη γέφυρα αυτή προς τους διάφορους άλλους τομείς. Η γέφυρα πρέπει να γίνει και προς την δομή των επιχειρήσεων εδώ θα παίξει ρόλο ο ρυθμιστής, σημαντικό ρόλο, καθώς επίσης θα παίξει σημαντικό ρόλο η διαφάνεια και η εποπτεία των χρηματικών ροών ή χρηματοδοτικών ροών, κάτι το οποίο ήταν κάπως θεωρητικό στο παρελθόν. Ωστόσο, χωρίς να λησμονούμε ένα πράγμα, δεν μπορούμε να μπερδεύουμε την παρέμβαση με οποιαδήποτε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού. Πρέπει να πούμε αυτές και αυτές οι δομές προκαλούν αδιαφάνεια. Αυτά πρέπει να τα κάνουμε τους επόμενους μήνες, ώστε από το σιδηροδρομικό πακέτο να βγει ένας παράγοντας πραγματικά ανάπτυξης και δημιουργίας απασχόλησης και να μην πάρει λάθος δρόμο. Σας ευχαριστώ. Λιμπεράτσκι, τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. ακολουθώντας ε, το πνεύμα του κυρίου Γκρός, δηλαδή μην θέλοντας να υιοθετήσω μια εξαιρετικά ριζοσπαστική άποψη και πάντοτε μεριμνώντας να πετύχουμε τους μακροοικονομικούς μας στόχους, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το 11%, το 11 των μεταφορών στην Ευρώπη γίνεται δια του σιδηροδρόμου. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να έχουμε ένα σύστημα μεταφορών διασυνοριακό που θα εκτείνεται σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πρέπει να αλληλοσυνδέονται και να λειτουργούν εύρυθμα μεταξύ τους τα εθνικά ε, συστήματα αλλά και τα περιφερειακά συστήματα. Οι επιβάτες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν και θα πρέπει οι δικές τους ανάγκες να λαμβάνονται υπόψη. Έχοντας λοιπόν αναλύσει όλα αυτά, στόχος μας είναι να επανέλθουμε σε αυτό το οποίο είχε πει ο Κοπέρνικος, ότι πολύ συχνά Άλλο είναι να χρησιμοποιούμε τα χρήματα και άλλο τα καλά χρήματα. Δηλαδή, ελήψη άλλων ε, επιλογών, συχνά οι επιβάτες χρησιμοποιούν τη χειρότερη δυνατή επιλογή. Η απελευθέρωση της αγοράς, η ιδιωτικοποίηση, ενδεχομένως είναι ένα μέσο για την επίτευξη του σωστού σκοπού, που είναι να έχουμε ένα σύστημα αποτελεσματικό. Δηλαδή, η απελευθέρωση της αγοράς, οι ιδιωτικοποιήσεις δεν πρέπει να γίνουν αυτός σκοπός. Η, άλλωστε η μεταφορά η δημόσια πρέπει να είναι προσβάσιμη, διαθέσιμη και από οικονομικής πλευράς για τον καταναλωτή αλλά και από κοινωνικής πλευράς και από άλλες πλευρές. Άρα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ορισμένες κοινωνικές προϋποθέσεις και κανόνες θα πρέπει να θέσουμε κατά μέρος επαρκή κονδύλια για όλα αυτά και θα πρέπει να το συζητήσουμε περαιτέρω. Να υπάρξει μεγαλύτερη διαβούλευση για το πόσα πολλά μπορούμε να διαθέσουμε για ένα δεδομένο δρομολόγιο ή για ένα δεδομένο τρένο. Να γίνουν υπολογισμοί αναεπιβάτη, αναχιλιομετρική απόσταση που διανύεται. Ε, εν πάση περιπτώσει, η δική μου εμπειρία στην Πολωνία με διδάσκει ότι οι διακονισμοί οργανώνονται με βάση το μειοδότη. Είναι πολύ πρακτικό αυτό. Το μόνο κριτήριο να είναι η τιμή. Και είναι και το καλύτερο παράδειγμα αυτού που έλεγα πριν. Πώς τα κακά χρήματα αντικαθιστούν τα καλά χρήματα. Ε, οι πιο σταθερές λύσεις δεν προτιμώνται πάντοτε δυστυχώς. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να θεσμοθετήσουμε επαρκή κριτήρια επιλογής, να έχουμε μια συνολική δέσμη, αυτή να είναι η προσέγγιση μας, να δεχθούμε ορισμένες υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Πάντοτε τίθεται θέματα για τον ΕΡΑ, ε, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνδυροδρόμων, αλλά και για τους εθνικούς οργανισμούς σιδηροδρόμων. Ε, πρέπει να δούμε ποιο είναι το καλύτερο για να έχουμε μια βιώσιμη σιδηροδρομική υπηρεσία. Είναι καλύτερο να κατακαιρματίσουμε την υποδομή ή μήπως είναι καλύτερο να εμείνουμε ε, σε μια προσέγγιση κοινοπραξίας και ε, συνολικής δράσης. Πολλά τα ερωτηματικά ε, και θα πρέπει να βρούμε τις τελικές απαντήσεις που θα καθορίσουν άλλωστε και τη μορφή που θα έχει το νέο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα. Να ξεκινήσουμε εκ του μηδενός και να το δημιουργήσουμε εξ αρχής. Ευχαριστώ κύριε Λιπεράτης και ο κύριος Τσιμός για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μετά την αδιατύπωση της τρίτης σιδηροδρομικής δέσμης. Μιλάμε τώρα για την τέταρτη σιδηροδρομική δέσμη, μας λέει ο κύριος Τρεμός, ή Cells. Και ελπίζουμε να έχουμε και αναδιατύπωση αυτού πριν φτάσουμε στο στάδιο της υλοποίησης και εφαρμογής. Αγαπητοί συνάδελφοι, να αναγνωρίσουμε ότι τα τελευταία δέκα χρόνια έχουμε εξετάσει τρεις σιδηροδρομικές δέσμες που στόχευαν να ανοίξουν τις εθνικές αγορές ώστε οι σιδηροδρόμοι, σιδηρόδρομοι να είναι πιο ανταγωνιστικοί. Όμως σήμερα το μοντέλο αυτό ε, υπάρχει σε, κάποια, σε κάποιες χώρες αλλά ε, καταραίει σε άλλες. Εγώ δεν είμαι κολλημένος. Ε, είμαι ανοιχτό στο να μάθω, να ακούσω άλλες απόψεις. Δεν υπερασπίζομαι τις ιδεολογικές μου γνώμες μέχρι τελικής πτώσεως, ούτε μπαίνω στη συζήτηση με διάφορα απριόρι ε, και ε, προκαταλήψεις. Ως προς την υποχρεωτική οργάνωση διαγωνισμού για την ανάθεση μιας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Δεν είμαι κατά. Είναι μια ιδέα που θα μπορούσε να στηρίξω. Εάν παραμείνουν τα πράγματα ως έχουν, δεν θα γίνει κανένας διαγωνισμός και άρα δεν θα υπάρξει καμία υπηρεσία που θα προσφερθεί. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε για ποιο μέγεθος ε, η προκήρυξη διαγωνισμού θα πρέπει να είναι υποχρεωτική. Να κάνουμε ανάλυση κόστους ωφέλεια σε επίπεδο ε, τοπικών δήμων για τη μεταβατική περίοδο πριν να γίνει υποχρεωτική η προκήρυξη διαγωνισμού. Δεν είμαι υπέρ μεταβατικής περίοδου. Γιατί, Γιατί έχουμε ήδη χάσει πάρα πολύ χρόνο. Και ε, δεν αλλάζουν τα σιδηροδρομικά με αρκετά γρήγορη ταχύτητα. Ως προς την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας και το άνοιγμα της αγοράς μπορούμε να βρούμε τρόπους να αποφύγουμε τις τρευλώσεις, να έχουμε σωστούς κανόνες και να έχουν όλοι πρόσβαση στην αγορά και να παρέχεται η δημόσια υπηρεσία. Όπως είπε και ο Φίλιπ Τεμπέικερ προηγουμένως, δεν πρέπει το επιχείρημα του ανοίγματο ε, της ανοιχτής πρόσβασης να επιτρέψει σε κράτη-μέλη να βασιστούν στον κανονισμό για την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας ώστε τελικά να εμποδίσουν νέες εταιρείε από το να μπουν στην αγορά. Χρειαζόμαστε ελάχιστες προϋποθέσεις και ελάχιστα πρότυπα για όλους. Ωστόσο, ένα παλαιό και δίσκαμπτο καθεστώς δεν μπορεί να διατηρηθεί ως έχει. Ναι, να σεβαστούμε τις συλλογικές συμβάσεις, ναι όμως ε, και στις ελάχιστες υπηρεσίες που θα πρέπει να προσφέρονται στον επιβάτη σε περίπτωση π.χ. απεργίας. Και αυτό το είχα πει στην διατύπωση της τρίτης δέσμης πριν από δύο χρόνια. Εγώ είμαι εισηγητής της σχετικής έκθεσης από πλευράς ανταγωνισμού ε, και ανταγωνιστικότητας. Υπάρχει σχετικό κεφάλαιο ε, για τους σιδηροδρόμους και η Κομισιόν έχει δημοσιεύσει πρόσφατα την ανακοίνωσή της. Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί στα θέματα κρατικών ενισχύσεων, στα θέματα παροχής παροχής ε, δημόσιας υπηρεσίας και στα θέματα διαφάνειας. Ευχαριστώ κύριο Συρίπη από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την τέταρτη δέσμη. Αυτή η διάθεση της Επιτροπής είναι ένας ανοιχτός συνδρομικός χώρος. Εκεί απασκοπούν όλες οι εκθέσεις ε, για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο αυτό. Τι γίνεται όμως. Να προσέξουμε πώς θα ανοίξει αυτή η αγορά και για την σχετική έκθεση υπάρχουν δύο θέματα τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η διάσταση η οποία αποδίδεται στο σεβασμό της αρμόδιας αρχής που έχει αναλάβει τις μεταφορές σε ένα χώρο, σε μια περιοχή. Δεν μπορούμε να τις επιβάλλουμε μια επιλογή. Είναι δική της επιλογή να περνάει μέσω μιας προκήρυξης διαγωνισμού είτε χέρι-χέρι να δίνει σε κάποιο πάροχο υπηρεσιών μια αγορά από τη στιγμή δε που σημειώνεται μια ικανοποίηση όσον αφορά το έργο το οποίο γίνεται από αστυνομικές πλευρές και των πελατών του συνόλου του κοινωνικού. Γιατί λοιπόν να αφισβητήσουμε τότε αυτή τη δυνατότητα αυτής της αρμόδιας αρχής της αποκαλούμενης από τη στιγμή που είναι θετικό το αποτέλεσμα. Και τώρα, αντίθετα, το πράγμα της Γαλλίας, χάρη σε αυτόν τον κανονισμό ο οποίος ισχύει αυτός ο κανισμός, ένας τοπικός φορέας θα μπορούσε να προκηρύξει ένα διαγωνισμό, να κάνει μια προκήρυξη για έναν ανταγωνισμό απέναντι στον ΣΕΦ που είναι ο κλασικός πάροχος, ενώ πρώτα δεν γινόταν αυτό το πράγμα στη Γαλλία, δεν ήταν δυνατό. Άρα λοιπόν μέσα της Ευρώπης να ξεκινήσει αυτή η δυνατότητα για τους τοπικούς φορείς, τις τοπικές αρχές, αυτό είναι κάτι που έχει τρομερή σημασία ανα, ε, προτείνει τώρα μέσω μια πρώτη προκήρυξη μια αρμόδια αρχή να γίνει κάτι τέτοιο. Από τη στιγμή που όλο ο κόσμο είναι ικανοποιημένο, ευχαριστημένο, νομίζω αυτό ξεπερνάει αυτό που θα πρέπει εμεί να επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη σήμερα να αναφέρω μια τρίτη διάσταση η οποία είναι η κοινωνική. Καθόλου μα καθόλου παρούσα δεν είναι στα πλαίσια αυτής της πρότασης αυτής της Επιτροπής. Νομίζω ότι θα πρέπει να επενεξεταστεί από εμά σαν βουλευτές. Δεν σημαίνει απορρίθμιση αγορά στο άνοιγμά τη, να δημιουργήσουμε dumping και να μειωθούν οι μισθοί. Δεν πρέπει να είναι αυτό ένα δόγμα. Μην νομίζουμε ότι θα υπάρξει μια καλύτερη προσφορά επειδή θα ανοίξει η αγορά. Όχι, δεν μπορούμε να την οθετήσουμε έτσι ότι θα είναι μια και έξω καταγεγραμμένη. Ενώ θέλουμε να είναι καρπημένοι όλοι, να είναι στην ώρα του τα τρένα, να υπάρχει μια ασφάλεια, μια υποδοχή, μια ποιότητα στις υπηρεσίες και οι τιμές να είναι καλές ώστε να μπορούν κατάλληλα να μετακινούνται οι ταξιδιώτες. Αυτό όλα μπορούν να γίνουν, πρέπει να γίνουν βάσει και του σεβασμού όλων αυτών των κοινωνικών Τυχών, που δεν υπάρχουν όμως στην πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει πάνω σε αυτές τις δύο πτυχές που έχουν τρομερή σημασία στην έκθεση USP να εργαστούμε πάνω σε αυτές μια δυνατότητα ελεγμών των αρμόδιων αρχών και μετά αυτό το κοινωνικό, αυτή η κοινωνική πτυχή διαφορετικά θα είναι μια δογματική, ένα δογματικό άνοιγμα της αγοράς θα προσφέρει εγγυήσεις για τις μεταφορές και θα απορριθμίσει από κοινωνικής πλευράς μόνο να πούμε αυτή την οργάνωση σε και από αστυνομική πλευρά στα διάφορα κράτη. Δεν είναι άλλωστε και ο στόχο που επιδιώκει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, περισσότερη και καλύτερη αστυνομική μεταφορά. Όχι όμως με παρόμοια πραγματική προσέγγιση. Περισσότερη ευληγησία και ευκαμψία, περισσότερη δυνατότητα ελεγμών για τις αρμόδιες αρχές. Σας ευχαριστώ. Ζέλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη γιατί έχω ήδη απαντήσει για την έκθεση του κυρίου Γκρός. Είχα ε, κάποιες σημειώσεις για τη διαχείριση του κυρίου Βλάσεκ και μπερδεύτηκα και δεν τις, είπα όταν, δεν τις διάβασα όταν συζητούσαμε το θέμα της διαχείρισης. Αλλά, εν πάση πτώση, έτσι εξοικονόμησα χρόνο του ή άλλως. Για σας κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, Μπράιν, για αυτό. Κύριε Βίλς, έχετε το λόγο. Ο κανονισμός PSO καταλήγει μετά από μια δεκαετία δύσκολης πορείας και τέθηκε σε ισχύ το 2009. Στην Γερμανία ο σχετικός νόμος μπήκε σε ισχύ από τις αρχές 13. Πριν τώρα εφαρμοστεί ο κανονισμός, ακόμη καλά καλά πάει να αναθεωρηθεί. Εγώ αυτό το θεωρώ λίαν αμφισβητήσιμο. Είμαι αντίθετη με τις προτινόμενες αλλαγές του κανονισμού. Η Κομισιόν είτε προσθέτει νέες επιβαρύνσεις ή προβαίνει σε τροποποιήσεις του περιθωρίου ελιγμών των αρχών απέναντι στο status quo. Και πάει να ρυθμίσει υποχρεωτικά τις ε, προσκλήσεις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, οι απευθείας αναθέσεις μπορούν να γίνουν το πολύ μέχρι τέλος του 2022, τιμή κατοφλίου κάτω από το οποίο μπορεί να γίνουν άμεσες αναθέσεις θα επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να μην κάνουν τις δημόσιες αναθέσεις εφόσον το κόστος είναι μικρό, είναι, δεν, ε, εφόσον το εξοικονομούμενο ε, ποσό είναι μέχρι το ύψος του ε, κόστους της ανάθεσης. Ορισμένοι παραπέμπουν στην εγγύηση της ελευθερίας επιλογής της δημόσιας αρχής. Αυτό δεν πρέπει να διατηρηθεί οπωσδήποτε. Αλλιώς το περιθώριο ελιγμών των τοπικών αρχών θα περιοριστεί ακόμη περισσότερο και πρέπει να φοβούμεθα ότι η ευρεία διαθεσιμότητα των υπηρεσιών των εγγύς σιδηροδρομικών συνδέσεων θα επιδεινωθεί. Απομένως θα έχουμε κοινωνικό ντάμπινγκ και σε βάρος των εργαζόμενων. Αυτά ευχαριστώ. Thank you, Mrs. Wills. Right, have a list of speakers. Ευχαριστώ κυρία Βίλς. Έχω ένα κατάλογο ομιλητών. Δύο λεπτά ο, καθ... ο καθένας. Mr. So, uh, Mr. Κύριε Χαντράουι, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ναι, δημιουργήθηκε μια σύγχυση που οφείλεται είναι συνδεδεμένες οι δύο εκθέσεις, ο Ματιέ και εγώ. Πάντως συμφωνούμε όσον αφορά την, τον προσανατολισμό. Σχετικά με την έκθεση εδώ, θα ήθελα να τονίσω κυρίως δύο σημεία. Και τα δύο σημεία αφορούν το ότι χρειάζεται μια κάποια ευληγησία και ευκαμψία, όπως το είπα, υπάρχει διαφορετική κατάσταση από το ένα κράτο στο άλλο. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα είναι ιδιαίτερα αυστηρή και άκαμπτη η νομοθεσία κυρίως όσον αφορά ρυθμίσεις που αφορούν μια κατάτμιση ακριβώς σε διάφορα σημεία και στις ε, συμφωνίες με το δημόσιο. Εδώ κάτι τέτοιο είναι απαράδεικτο απαιτείται ευκαμψία. Τώρα λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις συμφωνίες συμβόλαια. Όχι, αυτό είναι πολύ αυστηρό. Αυτό ισχύει και για το θέμα εάν όλες αυτές οι συμφωνίες πώς θα πρέπει να κλειστούν μέσω προκήρυξης κατάλληλης ή μήπως θα μπορούσε να υπάρξει μια απευθείας ανάθεση προβλέπει η Επιτροπή διάφορες δυνατότητες, αλλά υπάρχει μια αυκαμψία, επαναλαμβάνω λοιπόν, απαιτείται περισσότερη ευληγησία. Είναι δύο σημαντικά σημεία, τα οποία σίγουρα συνδέονται με όσα προηγουμένως είπα. Σχετικά με τον περιορισμό αυτής της αρχής της ανοιχτής αγοράς, όπως επίσης και την ανοιχτή πρόσβαση, το Open Access, αυτά τα πράγματα θα πρέπει να παραμείνουν σε σχέση μεταξύ τους. Ο κύριος Μπαχ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ούτε καν δύο λεπτά δεν θα χρειάζεται να μιλήσω. Είπα και προηγουμένως σχετικά με την επικουρικότητα. Το είπε και ο κύριος Τσιρουμπή ότι οι εθνικές αρχές οφείλουν να ε, μάλλον πρέπει να διατηρήσουν αυτό το δικαίωμα ανάμειξής τους και να γίνονται σωστά οι προκηρύξεις. Το γεγονός ότι δεν γίνεται πάντα έχει και σχέση με τις εδαφικές ιδιαιτερότητες και ενδεχομένως με ένα σιδηροδρομικό δίκτυο το οποίο λειτουργεί απόλυτα ικανοποιητικά για τους επιβάτες. Να, τώρα, να πάμε τώρα να καταστρέψουμε τα δίκτυα αυτά, αυτό δεν έχει κανένα νόημα και θα είναι και δαπανηρό και ο Ματιού Γκρός είπε πολύ σωστά ότι πρέπει να προσέχουμε ευλαβικά τα χρήματα των φορολογουμένων. Μην πάμε τώρα για λόγους ιδεολογικούς να κατακαιρματίσουμε δίκτυα τα οποία λειτουργούν μια χαρά. Και σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές συνθήκες αυτή είναι η συνήθιση πολιτική της Κομισιόν. Η Κομισιόν προωθεί τον ανταγωνισμό. Οι δε συνέπειες του ανταγωνισμού αυτού, όπως το κοινωνικό dumping, φορτώνονται στις πλάτες των χωρών μελών. Εδώ λοιπόν πάει να ανακατευθεί, ε, μάλλον εδώ, ε, εδώ μάλλον βρίσκω να λείπει μια ορθή αντιμετώπιση, ειδικά για τον ε, σιδηρόδρομο, τον τομέα του σιδηροδρόμου δηλαδή στην Ευρώπη. Ο κύριος Παγνιό για δύο λεπτά. και πρόεδρε, σε αυτό το τέταρτη δέσμη, για αυτή την οδηγία, νομίζω ήταν περισσότερο πολιτική. Σημαντικό είναι να τα συλλογιστούμε όλα αυτά, αλλά το σημερινό σύστημα με τη μορφή αυτή, όπως είπε και ο συνάδελφος πριν από λίγο, δεν φτάνουν στην ώρα του στα τρένα. Και σήμερα οι Ευρώπη οι χρήστες δεν είναι ευχαριστημένοι από το σύστημα. Αυτή η υπόσχεση για το άνοιγμα της αγοράς, ε, εντάξει, να μειωθεί το κόστος, να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών, όλα αυτά δεν ανταποκρίνονται, δεν καθρεφτίζονται, στην στην πραγματικότητα. Εδώ λοιπόν ε, πιστεύω ότι η πρώτη πρόταση της Επιτροπής, ε, αυτή η οποία είναι από την άλλη πλευρά από το 2019, δεν νομίζω ότι δημιουργεί αυτή την ισορροπία όπως, ε, όπως την επιθυμούμε. Αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα του ανοίγματο για τις δημόσιες υπηρεσίες ε, είναι έτσι ξαφνικά και απότομα. Το είδαμε και σε διάφορα κράτη-μέλη και μάλιστα τα τελευταία χρόνια. Σημαντικό είναι λοιπόν να μπορέσουμε να αντιδράσουμε και όχι να δημιουργήσουμε ένα ανταγωνισμό που να είναι εις βάρος της ποιότητας. Έτσι, ένα ανταγωνισμό που να μην είναι υπέρ του κοινωνικού ντάμπιν. Ήταν ένα ανταγωνισμό που να είναι εις βάρος της ασφάλειας. Όπως αυτό που έγινε στην Αγγλία τα τελευταία χρόνια Υπήρξαν διάφορες αρνητικές αντιδράσεις ε, κάθε φορά που αναφέρω το παράδειγμα αυτό. Πάντως βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αποδεσματικότητα, οικονομικές απώλειες τρομερές και ακόμα δεν υπάρχει καθόλου διαφάνεια. Έτσι μια ιδιωτική εταιρεία χωρίς μετόχους, στον ατάλογο σύστημα που το, από την άλλη μεριά το ανταγωνίζονται ε, επιδοτήσεις και ανταγωνισμός ακόμα προηγούμενα. Καταλαβαίνετε όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν ένα πρόβλημα, υπάρχει, δημιουργούν ένα πρόβλημα και όπως ε, το είπε και ο εκπρόσωπος των σοσιαλιστών και ο συνάδελφος Γκρός. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα κατάλληλο δρόμο για να περάσουμε από αυτόν, να πετύχουμε την ισορροπία και εγώ θα υποβάλει ορισμένες προτάσεις για να το πετύχω αυτό. Ο κύριος Μπισέτ για δύο λεπτά. Ναι κύριε Πρόεδρε προλή... Ο συνάδελφος Μάικελ Κράμερ ε, μας έκανε ένα λάθος ε, γιατί η κυρία Ιζαμπέλ Ντιράν σε τι αναφέρθηκε, στη διαχείριση και ξαφνικά εγώ που είμαι ο σκηδός συγητής της ομάδας ε, δεν μπόρεσα να πλάβω το λόγο για το θέμα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν να μπορέσω να παρεύω όπως το είχα προβλέψει τότε και που είχα τον αλλαγό χρόνο. Δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ δεν είχε στεγνώσει ακόμα το μελάνι της πρώτης συμφωνίας, το δεύτερο πακέτο πριν από τέσσερις μήνες. Και από τέσσερις μήνες τώρα είχαμε το χρόνο και συναντήσαμε πάρα πολλούς που ενέχονται σε αυτό, συζητήσαμε και με συναδεύους και με την Επιτροπή, με το Υπουργείο, με τους, με τους διαχειριστές, με τις επιχειρήσεις, με τους χρήστες. Πρώτα απ' όλα η προσέγγιση της Επιτροπής. Εγώ είμαι εισηγητή από την ομάδα για το κείμενο λοιπόν για την Επιτροπή. Τι λέει, ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν την επιλογή ανάμεσα σε δύο πρότυπα οργάνωση. Ουσιαστικά όμως ε, ο ίδιος έχει αυτή τη δυνατότητα να το κάνει. Πάντα το, για το ίδιο πρόκειται. Απλά αλλάζει το καπελάκι του. Και είτε με τη μια μορφή είτε με την άλλη. Εάν το κοιτάξουμε από πιο κοντά, αυτό το συνικό τείχος περιγράφεται τόσο λεπτομερακά που δεν βλέπουμε καμία διαφορά μέσα στις δυνατότητες. Α, λοιπόν δεν είναι και τόσο ειλικρινής αυτή η προσέγγιση. Αλλά και εκπλήσωμαι, το καταλαβαίνετε, έστω και αν δεν έχω απόλυτα επιστημονικά κριτήρια. Αλλά υπάρχουν ορισμένα πράγματα με επιχειρήματα, με μια ανάλυση του πώς επηρεάζουν τα πράγματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάμεσα στο σύστημα διαχείρισης και στο άνοιγμα στην ε, ε, και με τον ανταγωνισμό, αλλά αυτά δεν έχουν αποδειχθεί. Υπάρχουν μια στοιχεία πάντω τα οποία δεν τα βρήκα ακριβώ και για το πώ θα ξεχωρίζουν αυτά τα πράγματα σε θέματα ανταγωνισμού. Ορισμένα κράτη-μέλη δεν ε, παρουσιάζονται σε αυτού του υπολογισμού που θα άλλαζε κανονικά τα πράγματα με αυτέ τα νέα που υιοθετούνται. Και ε, εδώ επίση οι εμπορικέ μεταφορέ δεν λαμβάνονται υπόψη σε αυτή την κάθετη διαχωρισμό για την υποδομή και θα είχαμε εντελώ διαφορετικά αποτελέσματα. Δεν αποδεικνύει η ανάλυση αυτή ότι αυτή η αύξηση της ε, κίνησης ε, θα γίνει εις βάρος άλλων τρόπων μεταφορά. Ε, προσπαθεί να διακόψει ο πρόεδρος. Είπαμε δύο λεπτά, δύο λεπτά, δύο λεπτά και είσαστε δύο λεπτά και δευτερό λεπτά. Να αλλά διαθέτα τέσσερα λεπτά κανικά. Όχι, όχι, δεν, έκανα εγώ το λάθος. Το λάθος το έκανε η ομιλήτρια. Εγώ δίνω το χρόνο ομιλίας σε αυτή την επιτροπή. Στην ομάδα σας δόθηκαν τέσσερα λεπτά, η ομάδα σας μίλησε για τέσσερα λεπτά, τέλειωσε ο δικός σας χρόνος, εσείς μιλήσατε δύο λεπτά, επόμενη ομιλήτρια η κυρία Τζουγό για δύο λεπτά. Είμαι σύντομη. Διακόπτει ο προηγούμενος ομιλητής. Λοιπόν, Ακούσαμε μια κάποια άσκηση κριτική. είναι πολύ ρεσπαστικά τα μέτρα, το πρότυπο από ότι οι ίδιοι Βρετανοί που το διαπιστώνουν σήμερα ότι δημιουργεί προβλήματα για αυτό το θέμα. Σε αυτό που σκεφτούμε και ακούω από πάρα πολλού ομιλητέ ε, να μην έχουμε το ίδιο πρότυπο για όλου. Ε, υπάρχουν πολλά και διάφορα που ισχύουν σε επίπεδο Ευρώπη. Ε, εδώ έτσι ήρεμα σοφά να δούμε ακριβώ την τεχνική πτυχή όλων αυτών για την ασφάλεια, για το αέρα, το ένα το άλλο. Αυτή η δουλειά πρέπει να γίνει, χρησιμεύει αλλά ταυτόχρονα να μπορέσουν όλα αυτά τα πράγματα να επανέλθουν, να ζητήσουν την Επιτροπή, να επανεξετάσει, να αναθεωρήσει όλα αυτά μετά από τις σημερινές παρατηρήσεις έτσι ε, προς την επικουρικότητα πάμε και πάνω σε αυτά τα πράγματα τα οποία αμφισβητούνται ή που δεν είναι πλήρη για να μπορέσουμε να υπόψη μας τα σημερινά πρότυπα και να κάνουμε σήμερα πράγματα, να δούμε τις ειδικές συνθήκες στα μικρά κράτη, στα μεγάλα κράτη, τα μακρινά και τα πιο κοντινά και την κοινωνική πτυχή που είναι ανεπαρκή Νομίζω ότι υπάρχει πολύ δουλειά που πρέπει να γίνει από τεχνική πλευρά, Θα πρέπει να διαθέτουμε χρόνο για την διαχείριση αυτή, να μπορέσουμε να το προετοιμάσουμε και έτσι η Επιτροπή να επανέλθει με ένα καταλληλότερο και καλύτερα προσαρμοσμένο κείμενο. Αυτά λοιπόν υποβάλλω και σε εσά σαν πρόταση, όπω επίσης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Κράμαρ για δύο λεπτά. Είμαι κατά των μονοπωλίων, ό,τι μονοπόλια και να είναι, κρατικά ή ιδιωτικά. Αυτά δεν δέχονται καμιά επιρροή. Έχουμε τώρα και τις εμπειρίες μας από τον ανταγωνισμό, όπου υπάρχουν και αρνητικές επιπτώσεις και θετικές. Όταν ανοίξαμε το πακέτο της μεταφοράς εμπορευμάτων, ορισμένες χώρες μέλη άνοιξαν τις ε, μεταφορές εμπορευμάτων, είδαν να αυξάνονται οι μεταφορές τους, 36% ορισμένες. Η Γαλλία τα κράτησε κλειστά Μείωση 27%. Χάνονται δουλειές, χάνεται η οικονομία. Έρχομαι τώρα σε ένα άλλο. Düsseldorf Cast Μέτμαν. Επρόκειτο να την κλείσει ο σιδηρόδρομος διότι τη χρησιμοποιούσαν 500 επιβάτες. Τώρα, 12 χρόνια μετά, έχουμε φτάσει σε 23.000 επιβάτες. Το άνοιγμα δηλαδή εκεί βοήθησε, διότι τότε ανοίχτηκε στον ανταγωνισμό η ε, γραμμή αυτή. Τώρα, η άμεση ανάθεση βεβαίως και πρέπει να είναι ελεύθερη. Δεν τρελαθήκαμε σε μια μικρή πόλη, μια επιχείρηση λεωφορείων με 10-12 γραμμές, να πάμε να κάνουμε πανευρωπαϊκή πρόσκληση ενδιαφερόντος. Ούτως ή άλλως μόνο 5% λαμβάνονται υπόψη πανευρωπαϊκά. Πρέπει ωστόσο να είναι δυνατό να γίνει και απευθείας ανάθεση. Όμως χρειάζεται και αμοιβαιότητα. Δεν είναι δυνατόν στη Γαλλία, στο Παρίσι, η ΕΡΑΤΕΠΕ να έχει την άμεση ανάθεση στη διάθεσή της για ένα τεράστιο έργο, ταυτόχρονα όμως να μπορεί να πάει στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα να πάρει το μετρό διότι εκεί πρέπει να είναι ε, προκήρυξη διαγωνισμού. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Πρέπει οι χώρες να αποφασίσουν. Δεν έχει καμιά σχέση αυτό με οποιαδήποτε δογματική τοποθέτηση. Όταν μια επιχείρηση χέρι της δυνατότητες άμεσης ανάθεσης, αυτό ισχύει και για τις θηγατρικές του, δεν μπορεί μετά να έχει διπρόσωπο παιχνίδι και να κάνει και άλλα. Ευχαριστώ. Προχωρούμε τώρα στον κανονισμό που ανακαλεί τον κανονισμό 1192. Ελπίζω να μην χρειαστούμε πολύ χρόνο Κυρία Βίλς, θα κάνετε την εισαγωγή εξ ονόματος του κυρίου Κόλιτσεκ. Παρακαλώ να είστε σύντομοι, όσο πιο σύντομοι μπορείτε. Ο Κόλιτσεκ δεν είναι παρόν σήμερα, γι' αυτό θα πω τώρα κάτι για τη θέση του εισηγητού. Η Κομισιόν προτείνει ο κανονισμός 1129-69 ε, να αρθεί μέσα στα πλαίσια του πακέτου των σιδηροδρόμων. Ο κανονισμός αυτός έχει επιτρέψει στις χώρες μέλη μέχρι τώρα να υποστηρίζουν χρηματοδοτικά ορισμένες σιδηροδρομικές εταιρείες που, για να αντιμετωπίσουν πάνες που δεν έχουν άλλοι, άλλοι τρόποι μεταφορών. Εκεί χωρίζονται σε 15 διαφορετικές κατηγορίες. Για παράδειγμα, συνταξιοδοτικά για τους σιδηροδρομικούς, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται νωρίτερα από ε, άλλες κατηγορίες, Επίσης για ορισμένες διασταυρώσεις. Ο κανονισμός είναι ε, χρονολογείται ακόμα από την εποχή των εθνικών σιδηροδρόμων και γι' αυτό περιλαμβάνεται ονομαστικός κατάλογος των εταιριών αυτών. Έχει προσαρμοστεί βέβαια το ε, τελευταία το 2007 και περιλαμβάνει τώρα 36 συνολικά επιχειρήσεις. Τέσσερις μόνο χώρες μέλη Βέλγιο, Γερμανία, Ιρλανδία και Πολωνία έκαναν χρήση αυτή τη δυνατότητα. Η Κομισιόν θεωρεί ότι ο κανονισμό δεν προσαρμόζεται πλέον με τη σημερινή νομοθετική πραγματικότητα και πλέον αυτού ε, προβαίνει και σε διακρίσει. Αυτό το τελευταίο σίγουρα είναι αληθέ. Συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο 36 ε, επιχειρήσεις μπόρεσαν να υποφεληθούν από κρατικέ επιχορηγήσεις. Επομένως αυτό δεν ε, εξασφαλίζει καμιά ισορροπία. Ο εισηγητής ωστόσο θεωρεί ότι είναι πρόωρο ακόμα να καταργηθεί η δυνατότητα τέτοιων ενισχύσεων. Ο εισηγητής προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανέλθει το 2017 με έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού στις επιμέρους χώρες μέλη και να συνοδεύεται αυτό από μια αξιολόγηση του κόστους και αυτό να το απευθύνει στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Τέτοια έκθεση θα επιτρέψει να δούμε εάν είναι απαραίτητο να αναδιατυπωθεί ο κανονισμός ή να αρθεί, να καταργηθεί. Οι χώρες μέλη καλούνται να να ε, εφαρμόσουν τον κανονισμό μέχρι 16 Ιουνίου 2015. Στο δε άρθρο 15 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει αναδιετία έκθεση στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την ε, εποπτεία και κατάσταση αγοράς. Η πρόταση να ληφθεί ως έτος αναφορά το 2017 είναι συνεπής, δύο χρόνια δηλαδή μετά από τη θέση της γη της, οδηγίας, της αναδιατυπωμένης οδηγίας. Με την έννοια αυτή θα κάνει και τις τροπολογίες του ο εισηγητής. Ο κ. Φέρμπερ δεν είναι παρόν. Α, δεν ξέρω αν το Λαϊκό Κόμμα θέλει κάτι να πει. Ο κ. Πανιού, θέλετε εσείς να πείτε κάτι. Σύντομα, σύντομα. Αυτή, αυτό εδώ, τι κάνει στα κρατημέλη, του επιβάλλει να βοηθήσουν ε, ε, για τη σύνταξη αυτών των εργαζόμενων ε, Εντάξει, θα μπορούσαμε να είμαστε ε, νέοι όχι για αυτή την κατάργηση, αλλά θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς, πώς επηρεάζουν τα πράγματα για το καθεστώς στο συνδεθεωτικό. Μας λέει η Επιτροπή ότι η κατάργηση αυτή στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ίσα ίσα που θα επηρεάσει σχετικά με αυτό, αλλά δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να ζητήσουμε μήπως ε, στα κράτη-μέλη, σε εθνικό επίπεδο, να δούμε, να ζητήσουμε μια εκτίμηση όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γαλλία. Διαφορετικά, έτσι, προκαταβατικά ξεκινώντας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά θα πρέπει όμως να υπάρξει ένας κάποιος έλεγχος, μια επελήθευση σε επίπεδο κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τρεμόσα, θέλετε να το σχολιάσετε? Όχι, τότε πάω στον κύριο Σιρήπη για τους πρασίνους. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Και εγώ εντάσσομαι ε, στη σειρά των ομιλητών που συμφωνούν με τον κύριο Παχνιό. Δεν υπάρχει αντίθεση. Μπορούμε όλα τα κράτη-μέλη να τα βάλουμε στο ίδιο επίπεδο. Όλοι να παίζουν βάση των ίδιων κανόνων. Δεν θα είναι σημείο τριβής κατά τη γνώμη μου. Θα βρούμε συνένεση πιστεύω και μάλιστα σχετικά εύκολα. Ο πρόεδρος για την Επιτροπή, η κυρία Γιάγκερ.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 Εξ ονόματος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μάθιου Γκρός γιατί μας υπενθύμησε ότι η Κομισιόν προσκλήθηκε στις διαπραγματεύσεις για την αναδιατύπωση και υποβάλαμε πρόταση για το άνοιγμα της εγχώριας αγοράς και για την επιβολή ανεξάρτητων διαχειριστών υποδομών. Ασκείται κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί υποτίθεται δεν παρέδωσε το παραδοτέο. Όμως με χαρά μου βλέπω και θα αναφέρω στους ανωτέρους μου ότι ε, σχεδόν εμπρόθεσμα καταφέραμε να παραδώσουμε τα παραδοτέα κατά γενική ομολογία σε αυτήν εδώ την Επιτροπή κατά τη διάρκεια του 2013. Κανείς δεν είπε ότι θα ήταν εύκολο το άνοιγμα μιας εγχώριας αγοράς από τη στιγμή που το 94% της μεταφοράς επιβατών για τη συνδροδρομική οδού γίνεται στην εχώρια αγορά και γι' αυτό θεωρούσαμε ότι η πρόκληση ήταν πολύ μεγάλη. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες από τις ανησυχίες σας και να τις καταλαγιάσω. Ο κύριος Ζήλια έθεσε ερώτημα για το τι επιθυμούν οι πολίτες μας. Το Ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν το άνοιγμα της αγοράς για να έχουν υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών. Η κυρία, ο κύριος Ντεμπέκερ λέει ότι το άνοιγμα της αγοράς από μόνο του δεν αρκεί, καθώς ε, τα δύο τρίτα των σιδηροδρομικών υπηρεσιών εντάσσονται στο κανονισμό για την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Άρα αυτά ε, πρέπει να συνάδουν με υποχρεωτική προκήρυξη διαγωνισμού για την ε, ε, παροχή δημόσιας υπηρεσίας και άρα πρέπει να μεταρρυθμιστεί και να αναθεωρηθεί ο σχετικός κανονισμός. Κύριε Ζηρήπη, να σας πω ότι το άνοιγμα της αγοράς δεν σημαίνει ανεξέλεκτη απελευθέρωση ή ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρομικών υπηρεσιών. Θα προτείνουμε πολύ λεπτομερείς κανόνες για το πώς θα γίνουν όλα αυτά. Θέλουμε να αποφύγουμε ε, το à la carte, το να διαλέγει κανείς μόνο ό,τι του αρέσει οι εταιρείε να ε, ξεκινούν νέες υπηρεσίες στις πιο κερδοφόρες γραμμές, αλλά αυτό το θέλουμε, αλλά θέλουμε να διασφαλίζεται και η δημόσια υπηρεσία ταυτοχρόνως. Θα πρέπει να υπάρξει οικονομική ισορροπία, να γίνει τεστ γι' αυτό και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα αναλάβουν αυτή την υποχρέωση, να κάνουν αυτά τα τεστ, αυτές τις δοκιμές για που θα επιβεβαιώσουν κατά πόσο υπάρχει σωστό σημείο ισορροπίας. Και εδώ απαντώ στον κύριο Ελχαντράουι. Στον κύριο Κράμερα απαντώ λέγοντας ότι εμείς θεωρούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισμών θα πρέπει να είναι ο κανόνας. Ωστόσο, ο κανονισμός προβλέπει εξαιρέσεις. Επιτρέπει την απευθείας ανάθεση όταν τα κριτήρια είναι σαφή και αντικειμενικά. Και σίγουρα συμφωνείτε με αυτό, έτσι δεν είναι, κυρίως με τον αντικειμενικό χαρακτήρα. Ως προς τον ορισμό της υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας και την ερώτηση του κύριου Μπαχ. Αυτό θα παραμείνει εντός της αρμοδιότητας των ε, σχετικών αρχών, ε, ρυθμιστικών αρχών. Είναι θέμα επικουρικότητας. Θα πρέπει να υπάρξουν ελάχιστοι κανόνες που θα διασφαλίζουν ότι η απόφαση, ε, η εκάστοτε πράξη να ενταχθεί στο κανονισμό PSO. Όταν γίνεται αυτό θα γίνεται βάση αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων για τα κατόφλια. Επίσης εφαρμόζουμε πλήρως και απαρεγκλήτως την επικουρικότητα Έχουμε τα προτινόμενα κατόφλια για τα χιλιόμετρα και για την δημόσια υπηρεσία σε κράτη-μέλη. Αυτό μπορεί να παρακινήσει τα μικρά κράτη-μέλη να επιταχύνουν την ολοκλήρωση. Η απάντηση είναι όχι. Υπάρχει αρκετή ευελιξία ως προς το σχετικό μέγεθος του κάθε ενός από τα τρία PSO. Πολλοί εξημών με ύψιλο λέτε ότι δεν θα ανοίξει η αγορά εάν δεν έχουμε παιχνίδι επί ίσης όρης. Η Επιτροπή δεν προτείνει υποχρεωτική αλλαγή. Και γιατί, θα σας το πω γιατί. Διότι η δομή, η διάρθρωση του σιδηροδρομικού κλάδου και τα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας των σιδηροδρόμων είναι τόσο διαφορετικά πράγματα από τη μία χώρα στην άλλη που ε, επιτάσσεται, είναι η ανάγκη να τηρήσουμε την αρχή της επικουρικότητας ώστε τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν ποια είναι τα πιο ε, κατάλληλα μέτρα προστασίας για το προσωπικό που εργάζεται εκεί, για το τροχαίο υλικό. Ε, ερώτηση του κυρίου Λιμπεράτσκι και κυρίας Τιουγό. Το άνοιγμα της αγοράς ε, δεν θα είναι αποτελεσματικό αν δεν αρθεί αυτό το τεχνικό εμπόδιο της πρόσβασης στο κατάλληλο τροχαίο υλικό. Αυτό είναι απαραίτητο, είναι ζωτική σημασία για να έχει επιτυχία ε, η διαδικασία του διαγωνισμού για την πιο ανταγωνιστική προσφορά. Έρχομαι τώρα στην αποσύνδεση, στην αποσύζευξη το άνοιγμα της αγοράς των επιβατών ε, θα πρέπει να γίνεται με πρόσβαση στην υποδομή με μη διακριτικό ή διακρισιακό ε, τρόπο, να μην γίνονται διακρίσεις. είτε και το δεύτερο αίτημα στην αναδιατύπωση. Θα επαναλάβω αυτό το οποίο ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριος Κάλλας, είπε. Εάν δώσετε τον έλεγχο των αυτοκινητοδρόμων σε μια εταιρεία φορτηγών δεν θα εκπλαγείτε τι θα συμβεί στους ανταγωνιστές της. Θα είναι βέβαιο το τι θα συμβεί στους ανταγωνιστές της. Έτσι δεν είναι. Θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι λοιπόν οι διαχειριστές των υποδομών, να είναι αποτελεσματικοί, άρα πρέπει να έχουν λειτουργική και οικονομική ανεξαρτησία και να υπάρχουν τα εχέγγυα της διαφάνειας για να μην πάμε μετά στα, ε, στη σύγκρουση συμφερόντων. Εσείς ζητάτε ενισχυμένη ανεξαρτησία και η Κομισιόν απαντάει λέγοντας ότι η θεσμική αποσύνδεση και αποσύζευξη του unbundling είναι η πιο απλή και πιο αποτελεσματική λύση γι' αυτό. Όσα κράτη-μέλη θέλουν να διατηρήσουν ενιαία δομή μπορούν να το κάνουν. Και αν επιλέξουν τέτοια άγουσα τότε πράγματι πρέπει να υψώσουν ένα ισχυρό στέρεο ε, συνικό τείχος για να διασφαλιστεί εκ των έσω η ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομών. Εμείς πιστεύουμε ότι η ισχυρή ρυθμιστική αρχή δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε και ανεξάρτητο διαχειριστή υποδομής. Ιδαλλιώς, οι εταιρείες που θέλουν να ξεκινήσουν να προσφέρουν υπηρεσίες σε μια χώρα όπου ελέγχουν τις υποδομές ε, θα πρέπει να ακολουθήσουν μακροχρόνιες και χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες δικαστικές και δικαστικής ματιαμάχες. Αυτό το έχουμε δει στο παρελθόν. Μιλήσατε και για το unbundling. Θα προσπαθήσω να απαντήσω και στο πρόεδρό σας, ο οποίος μας ε, ρώτησε για το κόστος. Ένα νούμερο, τα 6 δις κυκλοφορεί. Αναρωτιέμαι από πού προέκυψε. Δεν τεκμεριώνεται από πουθενά είναι στον αέρα το νούμερο αυτό. Γιατί να είναι τόσο ξεχωριστό να ξεχωρίσουμε το διαχειριστή υποδομών από την λειτουργία και την παροχή της υπηρεσίας. Ε, ε, θεσμική, από θεσμικής πλευράς είναι κάτι που γίνεται ήδη. Δεν πιστεύουμε ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Η ανάγκη ύπαρξη συνικού τείχους. Συμφωνώ με τον κύριο Κράμερ δεν είναι αποδεκτό τα χρήματα του φορολογουμένου που προορίζονται για υποδομή να μεταβιβάζονται και να εμβάζονται σε άκαμπτους φορείς εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων οι οποίοι θα τα χρησιμοποιούν για οποιοδήποτε σκοπό. Όχι, πρέπει να πηγαίνουν στις υποδομές τα χρήματα αυτά. Και έτσι θα διασφαλίζεται η οικονομική και χρηματοδοτική διαφάνεια. Μπορώ να προχωρήσω αναφέροντας ε, και τις ρήτρες της επαλήθευσης και όλα αυτά. Επειδή όμως έχω μόνο ένα λεπτό στη διάθεσή μου, θα πω το εξής. Φεύγει η νόρμα, ο κανόνας για την τυποποίηση των λογαριασμών για τα θέματα αυτά και καλώς γιατί είναι αποξιωμένο. Ήταν ένας κανόνας που είχε υιοθετηθεί όταν δεν υπήρχε εσωτερική αγορά και όπου τα μονοπόλια βασίλευαν. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να ισχύει κάτι τέτοιο πλέον και καλώς διαγράφεται αυτός ο κανόνας. Στο κύριο Γκρός λέω ότι χθε υιοθετήσαμε τις ειδικέ συστάσεις ανά χώρα για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και θα δείτε πολλά στοιχεία που συνδέονται με τους σιδηροδρόμους. Η τέταρτη δέσμη σιδηρόδρομων είναι εξαιρετικά σημαντική για την ανάπτυξη ανάπτυξη για τις θέσεις απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια. Θα είναι μεγάλη χαρά για εμάς να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί σας με το Συμβούλιο και με το Κοινοβούλιο για την εύρυθμη υιοθέτηση της τέταρτης δέσμης σιδηροδρόμων. Σας ευχαριστώ και ελπίζω ότι τήρησα το χρονοδιάγραμμα. Ο Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ πράγματι τηρήσατε το χρόνο που σας είχε δοθεί. Δύο λεπτά σε κάθε εισηγητή, παρακαλώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πρωτίστως τους συναδέλφους και τις συναδέλφους για τις παρεμβάσεις των. Θα τα λάβω υπόψη. Θα συναντήσω βέβαια και προσωπικά τις επόμενες ημέρες τους και συγητές σχετικά με τα όσα είπε η Κομισιόν. Βέβαια, κατανοώ ότι η Κομισιόν επιθυμεί να υποστηρίξει την πρότασή της. Δεν την μέμφωμαι γι' αυτό. Ωστόσο, όποιος ισχυρίζεται ότι η απελευθέρωση έχει μόνο καλές πλευρές πρέπει να είναι λίγο προσεκτικός γιατί δεν είναι δεδομένο αυτό. Εμείς θέλουμε να επιτύχουμε τον στόχο μας. Ο στόχος μας συνίσταται στο να υπάρχουν ποιοτικές υπηρεσίες για τους επιβάτες. Από την άλλη μεριά χρειαζόμαστε κάποια ευελιξία. Χρειαζόμαστε κάποια οικονομικά κίνητρα μέσα στο σύστημα, χωρίς ωστόσο να υπερβούμε κάποια όρια που κινδυνεύουν να οδηγήσουν στην επιδίνωση της ποιότητας της προσφοράς. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή νομίζω και σε άλλο χρονικό σημείο. Εσείς κύριε Γκρός τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τις και τους συναδέλφους. Βεβαίω θα συνεχίσω και εγώ τη συζήτηση με τους Σκιώδης και με τους συναδέλφους εκείνους οι οποίοι επιθυμούν να συμβάλλουν. Απατώντας την Κομισιόν, νομίζω καλώς έπραξε να μας θυμίσει αυτά που είχαμε ζητήσει, αλλά σήμερα λέμε στην Κομισιόν ότι χρειαζόμαστε και περισσότερη ευελιξία σε ορισμένους τομείς και ελπίζω να παραμείνει το ανοιχτό πνεύμα της Κομισιόν, ότι δηλαδή η ανάθεση πρέπει να γίνεται για παράδειγμα ε, στη βάση του κριτηρίου της αποτελεσματικότητας. Υπενθυμίζω επίσης κάτι που είναι σημαντικό για μένα. Είμαι πεισμένος ότι εάν συγκεντρώσουμε διακομματικά όλες τις δυνάμεις που επιθυμούν να προωθήσουν την ε, πρόταση, τότε λέω αύριο ο σιδηρόδρομος μπορεί να γίνει το νέο Airbus για την Ευρώπη. Αλλιώς θα χάσουμε μια τεράστια ευκαιρία και για την έρευνα και για την κινητικότητα και για την απασχόληση. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση στα μάτια μου. Και σε αυτό θα μετρηθεί η προσπάθειά μας. Αυτή λοιπόν θα είναι η πρότασή μας, όχι μόνο προς την Κομισιόν, αλλά και συνολικότερα από τη δική μας Επιτροπή προς το Συμβούλιο Υπουργών, που είναι ο βασικότερος συνομιλητής μας και τον οποίο, και τον οποίο οφείλουμε να πείσουμε να εγκαταλείψει τα εθνικά όρια του σκέπτεστε και να προχωρήσει σε μια ευρωπαϊκή λύση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι ε, ο κ. Κόλτσεκ δεν είναι παρόν και η κυρία Βίλς δεν είναι σε θέση βέβαια να συνοψίσει την άποψή του. Ευχαριστώ λοιπόν όλες και όλους που επιμείνατε ότι πρέπει να σκεφτόμαστε πανευρωπαϊκά. Αυτό είναι σημαντικό. Να πω τώρα σε όλες και όλους ευχαριστώ. Σας υπενθυμίζω ότι η επομένη συνεδρίαση θα γίνει Δευτέρα 17 Ιουνίου στις 3 το απόγευμα. Και ευχαριστεί ο Πρόεδρος και τους διερμηνείς για την προσπάθειά τους. Οι διερμηνείς ευχαριστούν τον Πρόεδρο.